Buenas tardes. Καλό σας απόγευμα σε όλους. Καλό σας απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε. Στο σημείο της ημερησίας διάταξης αφορά την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Σας προτείνω να εθετήσουμε την εξή αλλαγή για την ημερησία διδαξή Σημείο 9. Η έκθεση του κ. Καλιού για την επέκταση Σέγγεν στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Θα συζητηθεί όταν καταφτάσει ο συγητής, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη διακοπή των πτήσεων. Και το σημείο 10, πρόσβαση στα έγγραφα. προτείνω να αναβληθεί για να συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση ΛΥΜΠΕ, προκειμένου να έχουμε διαθέσιμη, διαθέσιμο το σχέδιο της έκθεσης σε όλες τις γλώσσες. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι κρίνουμε την ημερησία διάταξη με τις αλλαγές αυτές και περνάμε στο σημείο 2 ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Καταρχήν, να σας εκφράσω την ικανοποίησή μου για το αποτέλεσμα της ε, πρόσφατης ε, επίσκεψης της αντιπροσωπείας ΛΕΜΠΕΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η έκθεση θα σας ταλεί σύντομα. Είχαμε μία σειρά επικοδομητικών συζητήσεων και νομίζω ότι το έργο μας θα καταστήσει δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θετήσει σημαντικό ψήφισμα. Όλοι θεωρούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στην Ολομέλεια. Την περασμένη εβδομάδα. Και όπως γνωρίζετε, ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Μελλοντικής Συμφωνίας TFTP θα λάβει η χώρα σήμερα και αύριο. Ο κ. Ράιχαν Πρι, διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 12 Μαΐου θα ενημερώσει τις πολιτικές ομάδες για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων για την TFTP. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το όλο αυτό το θέμα με την Επίτροπο Μάλστρομ. Αλλά και σε μελλοντικέ συνεδριάσεις. Τώρα. Α περάσουμε στο σημείο 3. Παρουσίαση από την Επίτροπο Μάλστρομ των πρόσφατων και τραχουσών εργασιών της Επιτροπής στον τομέα των αρμοδιοτήτων της από τη στιγμή τη ένδειξη τη αιτίας τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπός Μάλστρομ ζήτησε να έρθει εδώ στην Επιτροπή μα και να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για πρόσφατα ζητήματα που απτονται των αρμοδιοτήτων τη. Είμαστε πρόθυμοι να την ακούσουμε και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παρεμβάσεις και ανταλλαγή απόψεων. Κυρία Μάλστρομ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, αν και σας έχω συναντήσει ορισμένους εξημών σε άλλα βήματα και είναι η πρώτη φορά που συναντώ την Επιτροπή από την έναρξη της ε, θητείας μου, από την ακρόαση. Και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε τακτικά και σε αυτό το βήμα. Ξέρετε ότι έχει αναλάβει τα καθηκοντά τη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι εμεί, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προσπαθούμε τώρα να κατανοήσουμε πώ έχει νέα κατάσταση, πώ πρέπει να εφαρμόσουμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα και πώ πρέπει να συνεργαστούμε. Και φυσικά, ξέρετε, ω πλήρη συνομοθέτε, αναγνωρίζετε από όλου και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά και επικοδομητικά για τους τομείς που εντάσσονται στι δικέ μου αρμοδιότητε. και μάλιστα είναι η στιγμή όλα τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εστιάσουν τώρα στην ουσία των θεμάτων και να δώσουν λιγότερη προσοχή στα τυπικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που ε, εντάσσονται στον τομέα ΔΕΗ και ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τι έχει υλοποιηθεί, τι προετοιμάζουμε και να σας πω και ποια είναι τα δύσκολα ζητήματα για τα οποία ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας στο μέλλον. Όπω ε, ξέρετε, η Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ και εγώ πριν λίγες εβδομάδε παρουσίασαμε το σχέδιο δράση για το πρόγραμμα τη Στοκόλμη, το οποίο θέτει ε, μια φιλόδοξη στρατηγική, μια φιλόδοξη ατζέντα για την εντολή. Και έχουμε πολλά να πράξουμε και φυσικά αυτό ε, συνάδει και με την απόφαση των Υπουργών που ελήφθη τον περισμένο Δεκέμβριο από τους Υπουργούς και επίσης ελπίζουμε να συνάδει και με τις επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών και με τις ανάγκες τους. Έχετε λάβει το σχέδιο δράσης, ελπίζω να είχατε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά και θα ήθελα να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας επ' αυτού είτε τώρα είτε σε μεταπίτα στάδιο. Το πρώτο μήνα τη εντολή μου, πριν τρει μήνε ανέλαβα τα καθήκοντά μου, παρουσίασα αρκετέ προτάσει. Χαίρομαι που τις παρουσίασα σε εσά, αλλά και στο κοινό. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλώ για το σχέδιο δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που παρουσίασα την περασμένη εβδομάδα και αυτό ενδιαφέρει όχι μόνο εσά ε, και το Συμβούλιο, αλλά και πάρα πολλέ μη καπαόμικρον για το πώ μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύπλοκο ζήτημα. Το σχέδιο δράση παρουσιάζει μια κοινή προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σεβόμαστε πλήρω τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και τη Χάρτα των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού το σχέδιο δράσης εντοπίζει κάποιους τομείς, κύριους τομείς δράσης, όπως η πρόληψη, τα περιφερειακά προγράμματα προστασίας, υποδοχή και ο εντοπισμός, η εξέβρεση βιώσιμων λύσεων. Και αυτά θελοποιηθούν με μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων που δεν περιορίζονται στη μεταναστευτική πολιτική, αλλά φυσικά αντιμετωπίζουμε και τις κυρίες οδούς ε, της μετανάστευσης και σε όλα αυτά υπερισχύει προστασία. Η Κομισιόν επίσης υιοθέτησε την πρώτη ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο η έκθεση προβαίνει σε μια αποτίμηση της πρόοδου της εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από την Γαλλική Προεδρία το 2008 και σε πώς εφαρμόζεται το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Σύλλου και παρουσιάζει συστάσεις για τα επόμενα έτη. Και καταλήγει στο συμπεράσμα ότι τα κράτη-μέλη έχουν κάνει κάποια πρόοδο, αλλά φυσικά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Μία από τις πρώτες προτάσεις που υλοποίησα έχει να κάνει και με προτάσεις που αφορούν την υπηρεσία Frontex, αναθεώρηση της εντολής Frontex για να δυναμώσουμε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, για να καταστήσουμε δυνατό να έχει Frontex το δικό της εξοπλισμό, τους δικούς της συνοριοφύλακες και να είναι πιο ανεξάρτητη σε ό,τι αφορά το συντονισμό των επιχειρήσεων. Η πρόταση επίσης στοχεύει στο να ενδυναμώσει την πτυχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όταν τα κράτη-μέλη θα έχουν ε, ουσιαστικά δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν σε μία επιχείρηση, αναγκάζονται να παραδώσουν ε, και να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά και τον εξοπλισμό αλλά και τη στελέχωση. Και θα το συζητήσουμε τον κύριο Μπουζουτήλ αυτό ο οποίο είναι αρμόδιο για το ΣΥΣ2 και το ΒΙΣ. Νομίζω ότι ε, το αξιότιμο όρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κ. Σκαέλιο, θα έχει καθυστερήσει λόγω ε, τη τέφρα. Και μπορώ να σα πω ότι έχουμε ε, κάποια συμπεράσματα της 23ης Απριλίου από το Συμβούλιο ΔΕΗ προς την κατεύθυνση αυτή σε σχέση με την εφαρμογή του Σέγγεν. Από τη σκοπιά της Κομισιόν θα παρουσιάσουμε ένα καθολικό πρόγραμμα με εκτιμήσεις του προπολογισμού στο Συμβούλιο σε δύο εβδομάδες, 3 και 4 Ιουνίου. Τώρα προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε, να τελειοποιήσουμε τις απαιτήσεις του συστήματος ε, μαζί με τις δοκιμές, μάλιστα δύο, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν το επόμενο φθινόπωρο. Και μόνο όταν γίνουν τα βήματα αυτά που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, να επιβεβαιώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου το πρόγραμμα και τον προπολογισμό. Και αν δεν είναι δυνατό αυτό, τον Οκτώβριο, μετά από το διάλειμμα των θερινών διακοπών. Για το VAS, ε, τα, ε, οι κυρίες δοκιμές του συστήματος ε, καθυστέρησαν το 2009 αλλά ξαναξεκίνησαν στις 6 Απριλίου φέτος. Είναι θετικά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα και η Κομισιόν έχει την πεποίθηση ότι ο κύριος Ανάγκοδος θα ολοκληρώσει το στάδιο των δοκιμών μέχρι την τέλη Μαΐου και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την Επιτροπή ενήμερη για όλα τα βήματα, για όλη τη διαδικασία με διαφανή τρόπο. Επίσης, Χαίρομαι που στα τέλη Μαρτίου μπορούσα να σας παρουσιάσω δύο προτάσεις ε, στην σημερινή νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Φυσικά όλα αυτά είναι τρομερά εγκλήματα που αλληλοσχετίζονται συχνά και πρέπει η απάντηση να είναι πολύ ισχυρή. Θέλουμε εδώ να έχουμε αυστηρότερες ποινές και ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε μια πρώτη εντελέχη απόψεων σε αυτήν την Επιτροπή και φυσικά ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σα και στο Συμβούλιο για να καταληξούμε σε συμπεράσματα. Να σα πω τώρα δύο για τις μελλοντικέ προτεραιότητες Καταρχήν για την ε, νόμιμη μετανάστευση, όπως ξέρετε, η παγκοσμιοποίηση παρέχει καλύτερες δυνατότητες για τους ανθρώπους ε, να ε, περνούν τα σύνορα. Υπάρχουν προκλήσεις που παρουσιάζονται από την αυξαμένη κινητικότητα των ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό δίκτυο διαχείρισης της μετανάστευσης. Επίσης γνωρίζουμε ότι η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μεγάλη συνεισφορά για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το καλοκαίρι, τι καλοκαιρινέ διακοπέ, θα σα παρουσιάσω δύο προτάσει για του επιχειρηματικού εργαζομένου και για ε, το ICT ε, γιατί προκειμένου να μπορούμε να διευκολύνουμε τη μεταφορά ε, κάποιων μετακίνηση με συγχωρείτε κάποιων εργαζομένων με δεξιότητες για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της μετανάστευσης, ε, ένας ε, στόχος που τόνισε στην ακρόση μου είναι ο εξή. Θέλω να ενδυναμώσω την ελληνική μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη πολλά μέτρα έχουν ληφθεί και έχουν υλοποιηθεί, αλλά κάποια κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ε, πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα συστήματα ασύλου του και πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ζήτησα από τι υπηρεσίε μου να εξετάσουν προσεκτικά τα αποτελέσματα του πιλωτικού προγράμματο για τη Μάλτα για ε, την επαναγκατάσταση όσων χαίρουν διεθνού προστασία και βάσει αυτή τη αξιολόγηση και τη εμπειρία θα αξιολογήσουμε τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα σε έναν πιο παγιωμένο μηχανισμό για τις θεωρήσεις. Όπως είπα στην ακροσή μου, η ανάλυση της ε, προόδου που έγιναν στην Βορσιορτσικοβίνη και στην ε, Αλβανία για το αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι μία από τις προτεραιότητες. Έχουμε εργαστεί ε, εντατικά στο θέμα αυτό και νομίζω ότι... Πριν δύο εβδομάδε στην Επιτροπή ενημερωθήκατε. Προετοιμάζονται τώρα νομοθετικέ προτάσει και ελπίζω να μπορέσω να σα τι παρουσιάσω σύντομα. Όπως επίσης είχαμε υποσχεθεί, τον Ιούλιο θα σας παρουσιάσω μια ανακοίνωση η οποία θα προβαίνει σε μια αποτίμηση των κύριων πολιτικών επιτευγμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θα τονίσω και ορισμένες κυρίες προκλήσεις. Στον τομέα αυτό είναι πολύ σημαντική η αποτίμηση. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει ζητήσει να το πράξουμε αυτό εδώ και καιρό και πρέπει να το πράξουμε. Ε, πριν να προτείνουμε νέα μέτρα, φυσικά η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, Κομισιόν ετοιμάζουμε μία ανακοίνωση για τη στρατηγική εσωτερική ασφάλειας που θα θετηθεί το φθινόπωρο θα βασίζεται στη στρατηγική που έχει οθετηθεί από το Συμβούλιο ΔΕΗ το Φεβρουάριο και θα συνάδει με το σχέδιο δράσης της Στοκχόλμης θα παρουσιάζει μία σειρά κοινών απειλών και θα αναφέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε αυτές τις απειλές, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς μπορούμε να υπερασπίσουμε τις αξίες μας και να σεβόμαστε ταυτόχρονα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πώς μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλα αυτά και φυσικά καλωσορίζω και τη δική σας συνεισφορά σε αυτό. Ο πρόεδρο ανέφερε το TFTP και τι σχετικέ συζητήσει. Ε, φυσικά, μόλι επιστρέψετε από τη Washington, ορισμένοι εξημών και, νομίζω, και ελπίζω να ε, ήταν επικοδομητικό το ταξίδι σα. Ε, φυσικό σημαίνει το ψήφισμα που θετήσατε την περασμένη εβδομάδα και συζητήσατε συζητήθηκε και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Δυστυχώ κάποιοι δεν μπορούσαν να περιβρεθούν λόγω των προβλημάτων με το ηφαίστειο και φυσικά έχω στενή συνεργασία με την συγγητρία και του σκιώδη συγγητή. Η εντολή του Συμβουλίου, που δεν έχει θετηθεί ακόμη επίσημα, γιατί υπήρξε επιφύλαξη βρετανική στο Κοινοβούλιο, δεν έχει οθετηθεί ακόμα. Ξεκινήσαμε όμως διερευνητικέ συζητήσεις με τους Αμερικανού. προκειμένου να ξεκινήσουμε επίσημε διαπραγματεύσεις το συντομότερο. Έχουμε φιλόδοξη ε, εντολή, θα είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσεις, αλλά φυσικά όπως ήδη παρουσιά... έχω υποσχεθεί είμαι έτοιμη να έλθω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας αναφέρω για τη σχετική πρόοδο. Επίσης, ε, ψηφίσατε και για το ψήφισμα για τα PNR, ταυτόχρονα με το ψήφισμα TFTP. Θα έχουμε μία ανακοίνωση για τη διαχείριση των πληροφοριών ε, στον τομέα GLS. Ε, αυτό θα είναι γενικό αναφέρεται σε όλα τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων που έχουμε, αλλά φυσικά το PNR, καταλόγιο δεδομένων επιβατών, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Νομίζω ότι έχει πολύ επικοδομητική στάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προτείνω ένα πακέτο σε εσά για τα PNR θα πρόκειται αρχικά για μια ανακοίνωση, για μια ε, εξωτερική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα PNR, στη συνέχεια δύο διαπραγματικές οδηγίες για, τη ε, διαπραγμάτευση με τις για τις συμφωνίες PNR με Αυστραλία και ΕΠΑ και στη συνέχεια ε, με τον Καναδά και τέταρτον μία νέα προσέγγιση και πρόταση για ένα ευρωπαϊκό PNR. Εργαζόμαστε σκληρά για τις πρωτοβουλίες αυτές, ελπίζω να τις παρουσιάσω σύντομα στην Κομισιόν και κατόπιν σε εσά. Και τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιους πολύπλοκους φακέλους ε, για τους οποίους θα πρέπει να συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες και αναφέρομαι κυρίως ε, σε όλο το πακέτο σύλλου και την πρόταση για την άδεια. Όπως ε, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που να είναι προστατευτικό, αποτελεσματικό και δίκαιο. Και θα είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Κομισιόν αυτό τα επόμενα έτη. Δεν είναι αποδεκτό στην Ευρώπη ε, όπου έχουμε τόσα πολλά κοινά στοιχεία ή δυνατότητε ε, να, να λάβει κάποιο άσυλο να ποικίλουν τόσο πολύ από χώρα σε χώρα. Και επίση δεν είναι αποδεκτό οι ετούντε ασύλου να τη χάνουν μεταχείριση. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν παρουσίασε προτάσει όπω γνωρίζετε ήδη εδώ και πολύ καιρό για την αναρμόνιση για, το, για την εναρμόνιση των μηχανισμών ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δώσουμε προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και στην αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του. Στι προτάσει αυτέ, επίση, είχαμε συμφωνία για το ΕΑΣΟ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξη Ασύλου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση αυτή και ευχαριστώ την κυρία Λάμπερτ για την εργασία τη. Αλλά κάποιε από τι προτάσει σε αυτό το πακέτο είναι πάρα πολύ δύσκολε, το γνωρίζετε και εγώ το γνωρίζω και νομίζω ότι κάθε στοιχείο του πακέτου ασύλου είναι ζωτικό στοιχείο του κοινού συστήματο ασύλου αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στα πλέον δύσκολα στοιχεία και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι μια συζήτηση που υλοποιώ με την επόμενη Βελγική Προεδρία και θέλω να την κάνω και με εσά και με τους ε, αρμόδιους συζητητές και σκιώδεις συζητητές για να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα σε κάποια από αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα. Και φυσικά καλωσορίζω προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τώρα την επανακατάσταση Πρόκειται φυσικά για ένα θέμα που σχετίζεται στενά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο για να βοηθήσει του πλέον ευάλωτου ε, πρόσφυγε και να επιμεριστεί τι ευθύνε για του πρόσφυγε με τρίτε χώρε. Στο πλαίσιο αυτό έχει προτείνει η Κομισιόν ένα κοινό πρόγραμμα επαναγκατάσταση και το θεωρούμε ω μια κύρια πρόταση για την ανάπτυξη τη εξωτερική διάσταση τη πολιτική ασύλου. Και λυπάμαι λοιπόν ε, που υπάρχουν αποκλήσει σε διαδικαστικά θέματα και εμποδίζουν την γρήγορη θέτηση τη πρόταση. Η πρόταση τη Κομισιόν είναι ένα πρώτο βήμα που επικεντρώνεται στην χρηματοοικονομική στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Πρόσφυγες βάσει της εμπειρίας ε, και της ε, παρουσίασης νέων πιο φιλόδοξων πρωτοβουλειών που προβλέπονται ήδη στο πρόγραμμα τη Στοκόλμη, Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια απόφαση για την ουσία τη πρόταση και να υιοθετήσουμε απλέ διαδικασίε για τι προτεραιότητε επαναγκατάσταση. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια υγιή χρηματοοικονομική διακήρυξη χωρί φυσικά να θέτουμε και σε κίνδυνο τη λειτουργία του Ταμείου για του Πρόσφυγε. Ταυτόχρονα βέβαια αν δεν βρούμε μια λύση ε, αυτοί οι οποίοι θα θυγούν τα μάλλα θα είναι οι ίδιοι πρόσφυγε. Και τέλος, ε, Πρόεδρε, για την πρόταση για την ενιαία άδεια είναι κάτι που αποτελεί τμήμα τη ε, στρατηγική μια συνολική ε, μεταναστευτική πολιτική τη Ευρώπη και έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο του προτινόμενη ε, οδηγία πλαίσιο να δημιουργείται μια ενιαία άδεια και που να αφορά την εργασία και την διαμονή είναι ένα κύριο στόχο τη Κομισιόν. Θέλω να εργαστώ μαζί σα για ένα ισορροπημένο κείμενο που θα καταλήξει σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε και η μεταχείριση ε, των υπηκών τροχωρών που έρχονται νόμιμα και διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να δώσω στου εποχιακού εργαζομένου, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, ένα ασφαλέ νομικό καθεστώ προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφαλειά του και φυσικά αυτό αιτιολογεί ειδική πρωτοβουλία από την Κομισιόν. Ελπίζω να τη στηρίξετε έτσι λοιπόν, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εξωτήμοι κύριοι βουλευτές, έχουμε φιλόδοξη ε, ατζέντα. Αυτό μόνο για τους επόμενους μήνες. Στο μέλλον θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας επικοδομητικά προκειμένου να προωθήσουμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική στρατηγική. Ευχαριστώ κύριε Μάρστρο. Ε, καταγράψαμε 20 ε, συναδέλφους που ζητούν τον λόγο πρέπει να βάλουμε χρονικά περιθώρια. Ο κύριος Κουέγιο που είναι ο εισηγητής για την επέκταση προς Βουλγαρία και Ρουμανία του Σέγγεν καθυστέρησε λόγω της τέφρας. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρες κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης για τη Ρουμανία και την ε, Βουλγαρία, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να προετοιμάσει τη γνωμοδότησή του. Επίσης, ε, ε, μου ζήτησε να τονίσω ότι ετήθηκε αυτή την πληροφορία από το Συμβούλιο, αλλά μέχρι τώρα τα έγγραφα δεν έφτασαν. Οπότε τώρα αρχίζουμε με τους συντονιστές τη συζήτηση και μετά θα ακολουθήσουν τα μέλη. Ο κύριος Μπουσουτήλ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μάλμστρομ που ήρθατε, μας διαθέσατε το χρόνο σας και μιλήσατε τόσο ειλικρινά. Ε, καταρχήν το πακέτο για το άσυλο. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το πακέτο για το άσυλο πριν από ένα χρόνο σχεδόν. Ένα χρόνο ήταν, γιατί σε 7 Μαΐου έγιναν αυτά. Είναι λοιπόν ένας χρόνος. Και οπωσδήποτε ε, δεν ε, καθυστερούμε εμείς. Όμως είναι σαφές ότι όταν ε, κάναμε, περάσαμε με πρώτη ανάγνωση θέσαμε σαφείς πολιτικές προτεραιότητες που δεν θέλουμε να τις εγκαταλείψουμε. Η αλληλεγγύη είναι το βασικό πολιτική προτεραιότητα και εννοούμε δηλαδή αλληλεγγύη τόσο με τους ετούντες άσυλο βέβαια, αλλά και αλληλεγγύη με τις χώρες που δέχονται τους περισσότερους ετούντες άσυλο και δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αυτή την εισρωή. Η πολιτική μας προτεραιότητα είναι σαφής λοιπόν και θα πρέπει να τύχει σεβασμό ανά πάσα στιγμή. Επίσης το πακέτο για το άσυλο. Χρήζει κάποια διευκρίνηση θεωρώ από σας. Γιατί από ό,τι κατάλαβα κάποια μέλη της Επιτροπής μας ε, πιστεύουν ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα στην πρότασή σας σχετικά με τους εποχικούς εργαζομένους και αυτό μπορεί να επηρεάσει και το χρονοδιάγραμμα του πακέτου για την άδεια. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να μας διευκρινίσετε πάλι. Ξέρω ότι το κάνατε, αλλά πείτε το πάλι έτσι καθαρά ότι εσείς θα υποβάλλετε πρόταση για τους εποχικούς πριν από το καλοκαίρι, γιατί η δήλωσή σας θα έχει αντίκτυπο το έργο της Επιτροπής μας για τον τοσχέτη της ενιαίας άδεια. Τώρα για το TFTP ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι το βασικό θέμα. Είναι η μεταφορά ε, πολλών μαζικών δηλαδή δεδομένων. Στην Ουάσιγκτον η Αμερικανική κυβέρνηση είναι ανοιχτή στις συνομιλίες συμπεριλαμβάνοντας και τα πιο δύσκολα θέματα όπως η μεταβίβαση δεδομένων μαζικά. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα είναι τι θεμελιώδεις πολιτικές αλλαγές είναι διατεθειμένη να εξετάσει η Κομισιόν, ούτως ώστε να λάβει πραγματικά υπόψη αυτό το βασικό εμπόδιο που έχουμε μπροστά μας και να το ξεπεράσουμε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές στην πολιτική της, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι διαβιβάσεις ε, ε, τέτοιου είδους ε, δεδομένων ή να περιοριστεί πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι απλώς θέμα να το κάνουν οι Αμερικανοί αυτό. Τέλος, για να ολοκληρώσω, εις ό,τι αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, μπορούμε να έχουμε σαφή θέση της Κομισιόν σχετικά με τον αποκλεισμό των δικτυακών τόπων. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό και δεν έχω καταλάβει αν η Κομισιόν θέλει να ε, αποκλείσει τέτοιου ιστοσελίδες ε, που έχουν παιδοφιλικό υλικό ή όχι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ όμως σας θυμίζω. Ε, το όριό μας είναι δύο λεπτά γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. κύριος Λαμπρινίδης. Χωρίς μικρόφωνο. Α, σας είμαι... Α, εσείς είστε συντονίστρια. Ναι, μάλιστα. Δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες στην κυρία Μάλψον. Για τους εποχικούς θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι αυτή η οδηγία με την ενιαία άδεια που ασχολείται κυρίως με αυτό. Και επίσης θεωρούμε κατεπήγον το θέμα αυτό. Επίσης το γενικό πλαίσιο για όλους τους ε, μετανάστες εργαζομένους από τρίτες χώρες. Πότε θα δώσετε ένα γενικό πλαίσιο ε, μετά από το εποχικό. Επίσης για το PNR Πότε σχεδιάζετε να δώσετε εντολή για διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Με το Καναδά, Αυστραλία, ΙΠΑ υπάρχουν. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία για τις διαπραγματεύσεις στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να έχετε υπόψη σας βέβαια πριν διαμορφωθεί πλήρωση εντολή. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση. Φαίνεται ότι αν αυτό είναι ο κατάλογος προτεραιοτήτων για τον επόμενο μήνα, να ρωτιέμαι τι θα πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Γιατί προφανώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολλές προτεραιότητες και εγώ δυσκολεύομαι να δω πώς θα ε, κατατάξω τις προτεραιότητες του καταλόγου. Πολύ σύντομα δύο ερωτήσεις γιατί και οι προηγούμενες ερωτήσεις αφορούσαν θέματα μετανάστευσης. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Επίσης, μιλάω για την επανεισδοχή και τις σχετικές συμφωνίες, ε, ιδιαίτερα με το Πακιστάν, τη σχετική συμφωνία. Ε, αλλά και με τη και Λιβύη έχουμε δύο παραδείγματα αυτά. Πώς μπορεί να διασφαλίσει η Κομισιόν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που θα σταλούν εκεί θα τύχουν σεβασμού. Αυτές οι χώρες πώς θα συμπεριφερθούν όταν θα υπάρχει καθεστώς διέλευσης ε, από άλλες χώρες. Η δημιουργία ενός Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή κάποιων θεσμικών οργάνων ή κάποιων διπλωματικών σωμάτων δεν ε, λύνει το θέμα. Και βέβαια μιλάμε για ανθρώπους εδώ και πρέπει να μας νοιάζει. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το μέλλον της του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Αν δω το πρόγραμμα δράσης της Στοκχόλμης, αναφέρει εκεί ότι θα βγει από το Eurojust, ε, ε, βγαίνει από το, το Eurojust στο μέλλον. Θέλω όμως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό ορίζοντα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα, τη διασυνοριακή εγκληματικότητα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε ε, ποινικά πρότυπα στην Ευρώπη ε, που θα προβλέπουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα των εναγωμένων. Φέτος και τα επόμενα χρόνια τι θα κάνετε εδώ και πόσο γρήγορα θα μας υποβάλλετε κάτι. Δηλαδή δραστηριότητες προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης Ευρωπαϊκού Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κ. Σάλμπρεχτ, ο επόμενος ομιλητής. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση σχετικά με τη Γενική Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων στη Διατλαντική Συνεργασία. Συγκεκριμένα, ποιο χρονοδιάγραμμα έχουμε. Με ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες. Με ενδιαφέρει να ξέρω πότε θα υπάρξουν οι πρώτες προτάσεις, πότε θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και πότε αναμένεται η έγκριση της, ε, του πακέτου σε συνάρτηση και με τις ε, διαπραγματεύσεις FTP και τη Συμφωνία PNR. Και η δεύτερη ερώτηση, μετά την αξιολόγηση των υφισταμένων μέτρων ασφαλείας, πότε θα γίνουν συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες και θα αναλυθούν μέτρα στα πλαίσια της αστυνομικής ε, συνεργασίας και ποια έχουν νόημα να συνεχιστούν από αυτά που ανακοινώθηκαν. Με ενδιαφέρει να μου πείτε πότε θα ληφθούν τα μέτρα αυτά. Και Και επίσης πότε ε, θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε, ε, κυρία, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε για το SWIFT. Νομίζω και ελπίζω ότι στις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα διεξάγεται θα υπάρχει θάρρος να παρουσιαστούν τολμηρές ιδέες για να αλλάξει σημαντικά η συμφωνία. Μετά Ανησυχώ λίγο μετά την που για την αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον, γιατί το σημείο κινήσεως των Ευρωπαίων είναι πολύ κοντά στο σημείο το τελικό των Αμερικανών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε νέες ε, ιδέες ε, στο switch θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ε, ξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και από τη δική μας την πλευρά και ε, τα δεδομένα μας να μην μεταφέρονται ε, ε, χωρίς συζήτηση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θέλει ένα ευρωπαϊκό κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Είναι γνωστό ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να βοηθήσει την Κομισιόν να κάνει lobbying υπέρ της ιδέας αυτής και εδώ και στις πολιτικές μας ομάδες ε, ψηφίσαμε υπέρ της επανεγκατάστασης. Εγκρίθηκε από το 95% ε, της Επιτροπής, των μελών της Επιτροπής. Οπότε και εμείς ανησυχούμε μην κολλήσουμε στα διαδικαστικά και τα διαδικαστικά είναι αυτές οι πράξεις κατεξουσιοδότηση, Ούτε η συγητές σου οι θα τις εφεύραν αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να ε, προχωρήσετε στην επανεκατάσταση που επηρεάζει πολύ και την εξωτερική πολιτική. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα καθαρά εφαρμοστικό μέτρο αυτό. Και όπως ε, μας ε, λέει και η νομική υπηρεσία εντάσσεται στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο διαφέρουμε, αλλά δεν πρέπει να κολλήσουμε λόγω αυτού. Και η Κομισιόν νομίζω ότι έχει, μπορεί να κάνει ε, ένα βήμα μπροστά και σε αυτή την περίπτωση θα συνεργαστούμε και εμείς για το θέμα αυτό της επανεγκατάστασης. Ο κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, μιλήσατε για την νόμιμη μετανάστευση. Θα ήθελα να μου πείτε αν γίνεται συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα σχετικά με την ανάγκη ή την αναγκαιότητα μιας μαζικής ε, μετανάστευσης. Ε, αναφέρεται τίποτα για την δυνατότητα απορρόφησης των νέων μεταναστών, λαμβάνεται υπόψη την ανεργία. Εδώ μιλάμε για 25 εκατομμύρια άνεργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί δηλαδή θα εγκαταληφθούν στη μοίρα τους για να ε, βρεθούν ε, φθηνότερες θέσεις εργασίας να προσφερθούν στους μετανάστες ή υπάρχει κάποια βραχυπρόθεσμη πολιτική που σχεδιάζεται. Και τι γίνεται με την ε, προσέλκυση ανθρώπων με ειδικότητες ειδικευμένων ή μιλάμε για ενειδικευτούς. Ο Λουί Μισελ ήταν υπέρ αυτή τη προσέγγιση όταν ήταν στην Επιτροπή, όταν ήταν Επίτροπο. Μια άλλη ερώτηση. Σχετικά με τις συμφωνίες επιστροφής με την Τουρκία, που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, η Τουρκία μας εφοδιάζει σταθερά και είναι και χώρα διέλευσης παράνομων μεταναστών. Και η Τουρκία εξέφρασε αντιρρήσεις σε μια τέτοια ιδέα συμφωνίας επιστροφής. Ε, σημειώθηκαν τίποτε εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, έχετε κάποια σχέδια μέσω πρόθεσμα. Λοιπόν, τέλος του πρώτου γύρου των παρεμβάσεων θα απαντήσει η κυρία Μάλμστρομ ή μήπως θέλετε να, ακούσετε, και, να ακούσετε και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Ας απαντήσω στον πρώτο γύρο, αν δεν σας πειράζει, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να... Ε, μπορεί να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις ε, μετά από αυτά που θα πω. Για τον κύριο Μπουσουτήλ, βεβαίω το πακέτο του ασύλου ε, ε, ε, σκόνταψε ο Συμβούλιο, όχι στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό Θέλω να σας ζητήσω και τη συμβουλή σας τι θα κάνουμε, γιατί πράγματι μπλοκαριστήκαμε και πρέπει να βρούμε λύσεις χωρίς να παρατηθούμε από τις προτεραιότητές μας και πράγματα που τα πιστεύουμε πολύ. Πώς θα προχωρήσουμε, γιατί πράγματι μπλοκαρίστηκε η κατάσταση και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό ούτε στην Κομισιόν ούτε στο Κοινοβούλιο. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε με δημιουργικές προτάσεις για τους εποχικούς εργαζομένους. Ναι, πριν από το καλοκαίρι, δεν ξέρω ακριβώς πότε, μάλλον τον Ιούνιο θα υπάρξει πρόταση. Για τις μαζικές διαβάσεις δεδομένων, πολύ το είπατε αυτό. Με το SWIFT, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, η ιδέα είναι να περιλαμβάνει και διαβίβαση τέτοιων δεδομένων. Κρίμα, αλλά τι να κάνουμε με την τωρινή με τον, συμφωνία δεν μπορούμε αυτό να το παρακάμψουμε. Πρέπει να βρεθεί κάτι καινούριο. Μπορεί, αλλά δεν γίνεται βραχυπρόθεσμα. πρόθεσμα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και κάτω είδαμε στις διαρευνητικές συνομιλίες με τους Αμερικανούς είναι να περιορίσουμε αυτά τα μαζικά δεδομένα που διαβιβάζονται ε, να είναι πιο στοχευμένα κάπως, να περιοριστούν και ήδη αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, δύσκολη η διαπραγμάτευση και περίπλοκη, αλλά αυτό έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε. Τώρα για τον αποκλεισμό του, των ιστοσελίδων με την στήριξη της Κομισιόν, αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν, συμφωνούν όλοι, δεν είναι μόνο δεν είναι δική μου ιδέα, είναι τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να κόβουν στην πηγή το παράνομο υλικό στο διαδίκτυο ε, αυτά τα πορνογραφικά, όλο το παράνομο υλικό θα πρέπει να αποκλείεται στην πηγή. Καμιά φορά αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο, γιατί είναι σε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η host και είναι πολύ δύσκολο. Καμιά φορά παίρνει πολύ χρόνο. Προτείνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη εκτός από το κλείσιμο στην πηγή να κάνουν όπως κάνουν 10-11 χώρες ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να συνεργάζονται με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με ε, την αστυνομία, για να μπλοκάρουν το πορνογραφικό παιδικό υλικό στο διαδίκτυο. Έχουμε όλες τις διασφαλίσεις, έχουμε όλες τις νομικές διαδικασίες που το επιτρέπουν. Δεν είναι γενικό μπλοκάρισμα του ίντερνετ, γιατί αυτό συζητήθηκε πολύ στη μπλογκόσφαιρα και σε ορισμένε χώρε. Πρόκειται για συγκεκριμένα ιστοσελίδε. και αυτό γίνεται ήδη 5-6 χρόνια τώρα σε αρκετέ χώρε. και θέλουμε να το επεκτείνουμε ω πρόσθετο μέτρο, γιατί βεβαίω το κλείσιμο είναι το πιο αποτελεσματικό. Θα επανέλθουμε. Η εποχική, ναι, κυρία Γκένς, θα υποβληθεί η πρόταση σε ένα γενικό πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες. Υπάρχει στο πρόγραμμα της Στοχόλμης. Θα συμπεριλαμβάνεται στην εντολή για το PNR με τις τρίτες χώρες. Ακόμα δεν τα έχω τα σχετικά κριτήρια. Θέλω να μιλήσω στην κυρία Ίντενβελτ, στην εισηγήτρια και στους σκιώδεις για αυτό το θέμα, γιατί ο στόχος είναι να έχουμε κοινά κριτήρια για όλες τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Και οι τελικές συμφωνίες μπορεί να διαφέρουν λίγο ανάλογα με τη χώρα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σειρά κοινών κριτηρίων αναλογικότητας, επικουρικότητας, πρόσβαση στα δεδομένα, προστασία κλπ. Και ελπίζω ότι σύντομα θα ε, διατυπωθούν όλα αυτά. Τώρα για την επανεισδοχή, η κυρία Βέμπερ και άλλοι έκαναν σχετική ερώτηση, μιλώντα για Πακιστάν κλπ. Βεβαίω, ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πυρηνικό ζήτημα. Υπάρχει ένα κεκτημένο διεθνού προστασία και επιστροφών. Στην οδηγία για τι επιστροφέ αυτό το θέμα τονίζεται ιδιαίτερα και κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί πριν γίνει εξατομικευμένη αξιολόγηση της κατάστασης του φακέλου του. Οπότε υπάρχει ισχυρή προστασία ενσωματωμένη στο σύστημά μας. Και αυτό είναι που ε, συζητούμε και με τους ομολόγους μας. Τώρα γιατί ο ε, εισαγγελέα. Είναι πολύ σημαντική πρόταση. Είναι η, πρόταση, είναι η ευθύνη του, της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ. μπορώ να το κοιτάξω για να σας απαντήσω τι χρονικό ορίζοντα έχει θέσει. Είναι περίπλοκο και στο Συμβούλιο το θέμα. Ε, είχε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά θα πρέπει να δω τις λεπτομέρειες και ευχαρίστως να σας ενημερώσω ή ε, το δικό της το καμπινέ. Κύριε Άλμπρεχτ, ναι, η, συμφωνία, η Γενική Συμφωνία Προστασίας Δεδομένων σύντομα μέσα σε ένα μήνα νομίζω θα εγκρίνει διαπραγματευτική εντολή κομισιών. Και αυτό είναι δουλειά της Αντιπρόεδρου Ρέντινγκ να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Και αυτό οπωσδήποτε θα πάρει κάποιο χρόνο αν θέλουμε να πετύχουμε διαπραγματεύσεις στο TFTP, αυτές θα είναι πιο μακροπρόθεσμες. Οι γενικότερες συζητήσεις εντάσσονται στις συζητήσεις αυτές επίσης. Εμείς θα εγκρίνουμε εντολή πριν από το καλοκαίρι και θα αρχίσουμε γρήγορα τις διαπραγματεύσεις. Προβλέπω όμως ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος, γιατί το σκοπός είναι να καλυφθεί όλη η γκάμα των ε, διαπραγματεύσεων με τους ε, Αμερικανούς. Η κυρία Ρέντινγκ αργότερα θα σας ενημερώσει περισσότερο γι' αυτά. Ε, ε πόσο κα, απαιτούνται τα δεδομένα ή το αργότερο 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει η αναθεώρηση. Πριν από το καλοκαίρι πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα και μετά το καλοκαίρι θα υποβληθεί η σχετική πρόταση για την διατήρηση των δεδομένων. Ε, για τα, ε, τις μαζικές αποστολές ε, διαβιβάσεις δεδομένων ε, είπαμε θα κάνουμε σκληρέ διαπραγματεύσει, αυτό θέλουμε. Έχουμε το σχέδιο εντολή από το Συμβούλιο, κάνουμε συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζω και συμμερίζομαι την αίσθηση αυτή που έχετε κι εσεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε κάτι, αλλά βέβαια ε, ανταλλάσσονται αυτά, μπορεί να περιοριστούν. Πάντω είναι μαζικέ διαβιβάσει. Μπορεί ο ορισμό να είναι πιο σκληρό, αυστηρό, αλλά οι Αμερικανοί δεν θα κάνουν πίσω πάνω σε αυτό το θέμα της, διαβίβασης, της δεδομένων. Τώρα για την επανεγκατάσταση. Ναι, δεν είναι σαφές ε, αυτές, αν είναι ας πούμε πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση. Αν ε, είναι, θα είναι πολύ επαχθής διαδικασία και ίσως είναι και αντιπαραγωγικό το σύστημα, γιατί δεν θα μπορούμε να κινούμε κινούμεθα γρήγορα στην επανεγκατάσταση. Ε, ελπίζω να βρεθεί καλή λύση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν ε, είμαστε πεπισμένοι εμείς ότι είναι η πράξη. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, για την όμιμη μετανάστευση, κύριε Κλάις, επίσης, αυτό που συζητούμε είναι, ότι, είναι το γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη χρειάζονται ε, εποχικούς μετανάστες, συνήθως στη Γεωργία. Βέβαια, η Κομισιόν οι Βρυξέλλε δεν πρόκειται να επιβάλλουν τίποτε. Αλλά αν τα κράτη-μέλη χρειάζονται εποχικού, θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, ούτω ώστε να μην υπάρχουν καταχρήσεις και να μην υπάρχει μαύρη αγορά. Τα κράτη-μέλη πάντω θα αποφασίζουν αν θέλουν νόμιμου μετανάστευση ή όχι. εμεί ε, απλώ θέτουμε το πλαίσιο για τους εποχικούς. Ε, αυτή θα είναι ανειδίκευτη βέβαια είναι αυτή. Ε, είχαμε την απόφαση για την μπλε κάρτα που θα, θα εφαρμοστεί του χρόνου. Ε, ε, αυτή είναι για τους ειδικευμένους. Είναι πολύ περιορισμένη η οδηγία και δεν ξέρω αν θα διευρυνθεί για να ληφθούν υπόψη και, άλλοι, και άλλες κατηγορίες, αλλά προς το παρόν αυτό έχουμε και για την επανεισδοχή με την Τουρκία. Με χαρά σας λέω ότι επιτελείται μεγάλη πρόοδος και πάμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και ήταν πολύ επικοδομητικοί οι Τούρκοι. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Και τώρα υπόλοιπο γύρος με τα υπόλοιπα μέλη. Παρακαλώ πολύ. Δύο λεπτά κατά μέγιστο. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις σκέψεις για το προβληματισμούς της κυρίας Μάρστρομ μόλις ακούσαμε κάθε πρόγραμμα δράσης απαιτεί οικονομικούς πόρους ε, συγκεκριμένους και σημαντικούς. Εξάλλου στην Επιτροπή μας ε, θα εξετάσουμε την πρώτη, πιθανότητα, την πρώτη δυνατότητα για τον προπολισμό του 2011 σχετικά με τα προγράμματα παρέμβαση. Τώρα, ουσιαστικά η ερώτησή μου έχει εξή. Τι θεωρεί η Κομισιόν ότι μπορεί να πράξει για το ζήτημα της, ε, των υπερπληθυσμών των φυλακών. Ξέρουμε ότι αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε ανθρώπινο ε, στους ανθρώπους, στους φυλακισμένους συγκεκριμένα και οδηγεί πολλές φορές ε, σε αυτοκτονίες. Όπως θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε κάτι για τους τοξικομανείς. Δεν θα ήθελα να αναφέρω πράγματα που έχουμε ήδη πει στο παρελθόν και κάτι ακόμα κάποια παραδείγματα για αυτή την ε, αλληλεγγύη η οποία απαιτείται σε ό,τι φορά την ε, ρύθμιση του προβλήματος της μετανάστευσης. Δηλαδή ποιες είναι οι συγκεκριμένε παρεμβάσεις ε, που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να κρατηθεί αυτή η αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να καταστεί πραγματικά υποχρεωτική. Εάν υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα σας ευχαριστώ. Κύριε Λαμπρινίδη το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα τρεις ερωτήσεις. Σχετικά με την ε, Τουρκία. Μερικές φορές είναι καλύτερο να μην ε, λέμε και να γράφουμε πράγματα, αλλά να αναλαμβάνουμε δράση. Και το κείμενο αναφέρει πως ε, Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μου δημιουργούν πρόβλημα. Στη σελίδα 6, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται πως Δυστυχώ μιλάει μακριά από το μικρόφωνο της Λαμπρινής και είναι δύσκολο να τον παρακολουθήσουμε. Από το κείμενό σας λοιπόν ε, ε, απουσιάζουν κάποια πράγματα. Ε, αυτό είναι το κείμενο εδώ που σας δείχνω. Σε αυτό αναφέρομαι. Μπορείτε λοιπόν να διευκρινίσετε όταν μιλάτε ότι διαπραγματεύσει πάνε πολύ καλά με την Τουρκία, εάν συμπεριλαμβάνετε και συμπληρώνουν τα άτομα τα οποία ε, διασχίζουν την Τουρκία και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και πρόσφατα από τρίτες χώρες, μιλάτε μόνο για Τούρκους οι οποίοι ε, φεύγουν και μεταβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσω καλύτερα αυτό το σύστημα σχετικά με την επικοδομητική στάση της ε, Τουρκίας τώρα. Να αναφερθώ σε μια ερώτηση που ετέθηκε προηγούμενη σε ένα, μια τροπολογία όλοι τονίσαμε την ιδιαίτερη σημασία για τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτήσει ένα δικό της μηχανισμό θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο μηχανισμός ε, για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα παρακολουθεί τι ακριβώ πράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η ερώτηση μου έχει εξή. Μπορείτε λοιπόν να ζητήσετε από τους Αμερικανούς τουλάχιστον αυτά τα οποία λαμβάνουν κάποιες δυτικές εταιρείε από το SWIFT. Και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ε, μήπως δεν μπορεί να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, ΗΠΑ, συγγνώμη, για αυτό το ζήτημα. Και τέλος, σε ό,τι φορά την ένταξη των μεταναστών, να, μπορείτε να μου πείτε εάν έχετε κατά νου κάποια συγκεκριμένα μέσα και τρόπους ένταξης των μεταναστών. Ε, προβλέπετε κάποια κονδύλια. Ευχαριστώ κύριε Λάτφορτ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καταρχήν να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικές δύο ανακοινώσει που δεν πολύ προσέχτηκαν. Ίσως δεν είναι το δικό σα τομέα, αλλά είναι πάλι κατά του ρατσισμού, αντισημιτισμού κλπ. Και ανησυχούμε πολύ που δεν πάνε καλύτερα τα πράγματα και με την ύφεση και τι οικονομικέ δυσκολίες μάλλον αναμένονται να δυσκολέψουν τα πράγματα. Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι η μάχη κατά τη διαφθορά. Αναφέρεται αυτό, αλλά είναι σοβαρό πρόβλημα δυστυχώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και εκτός αυτής. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Ε, περιμένω την έκθεση αξιολόγησης το πρόγραμμα των δικαιωμάτων ε, περάσπισης. Θα περάσει χρόνο μέχρι να έρθει όλο το πρόγραμμα και εντωμεταξύ υπάρχουν πολλά προβλήματα με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Συμπεριλαμβανομένων προβλήματα σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν ε, ζητείται η παράδοση ανθρώπων και πρέπει η Κομισιόν να δεχτεί ότι και να καταλάβει ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε ως θέματα. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, η ανακοίνωση για τη συλλογή πληροφοριών. Πρέπει επίσης να δούμε αν υπάρχει επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία θα περιμένουμε μέχρι το 2014 μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση για την αποτελεσματικότητα συνεργασίας αστυνομιών. Καμιά φορά υπάρχει η αίσθηση ότι αν βελτιωθεί η συνεργασία εκεί, γιατί πολλές φορές ε, λέμε ας πούμε ας βρούμε περισσότερα δεδομένα αντί να πούμε ας δουλέψει η αστυνομία πιο αποτελεσματικά με βάση αυτά που έχει ήδη. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Καταρχήν, στη συνομιλίες σας με την κυβέρνηση της Μάλτας μιλήσατε ε, και για την, μιλήσατε και για την ε, έξοδο ενδεχομένω από το Frontex. Επίσης, ε, η πορνογραφία και στο διαδίκτυο και πώς γίνεται το αποκλεισμό. Λέτε ότι το επιχειρείτε. Πώς αποδεικνύεται, αλλά γιατί εγώ δεν έχω δει απόδειξη ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, στο πρόγραμμα δράσης της Οκχόλμης, ε, πολλές προτάσεις έχουν ε, σχέση με την ανάπτυξη. Εσείς πώς διασφαλίζετε καλή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και πώς λαμβάνετε υπόψη η ανάπτυξη όταν ε, διατυπώνετε τις προτάσεις σας αυτές. Επίσης, στο πρόγραμμα δράσης της ε, Στοχόλμης ε, λέτε ότι μπορεί το, η Frontex να αναλάβει το ρόλο των εθνικών συνοριοφυλάκων. Αυτό πότε θα το ε, προτείνετε και πώς θα λειτουργήσει. Τέλος, επειδή τον, αν, ή μάλλον αν είναι τόσο σημαντικά για μας όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε γιατί δεν αναφέρονται στην Συμφωνία Επανεισδοχής με το Πακιστάν. Ε, ενώ αναφέρονται σε άλλες ε, συμφωνίες. Ευχαριστώ, κύριε Σπρόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μπαριστρόμ, περιέγραψε την ε, νόμιμη μετανάστευση ως όφελος προς όλα τα μέρη. Συνήθως ε, αυτό οδηγεί όλες τις χώρες ε, και του μετανάστες. Αυτό ισχύει κυρίως αν μαζική μετανάστευση λαμβάνει χώρα από χώρες ε, με χαμηλούς μισθούς σε χώρες με υψηλούς μισθούς ήδη. πρέπει κάποιες χώρες να δαπανίσουν για υποδομή, για στέγαση και μάλιστα ε, και οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν ε, και στερούν τις χώρες τους από τις δικές τους δεξιότητες. Ε, πολλές φορές οι χώρες θεωρούν ότι είναι μια ηθική πολιτική. Αυτό όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί τελικά οδηγούνται οι οικονομίες στο να τελματώσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, θέλουμε ε, δεν θέλουμε τελικά να υπάρχει στο τρίτο κόσμο ανεργία. Σε ό,τι αφορά το σε άσυλο θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η αναλογία που προέρχεται από τις όμορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από πολύ μακρύτερα και έχουν περάσει από πολλές χώρες μέχρι να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν έχουν περάσει την πρώτη ασφαλή χώρα τότε έχουν ε, τελικά ε, περάσει στη χώρα αυτή και θα πρέπει ε, να επιστραφούν στην πρώτη ασφαλή χώρα στην οποία έχουν περάσει αν όχι στη χώρα προέλευσής τους. Να ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ γρήγορα να περιγράψω το θέμα και να κάνω και κάποια ερώτηση. Βρισκόμαστε ενώπιον ενό ε, σχεδίου ε, δράση. Έχουμε το πρόγραμμα τη Στοκόλμη ε, και την εκπόνηση του σχεδίου δράση. Έχετε οκτώ σημεία τα οποία αναφέρονται σε πάρα πολύ ευρία θέματα όπω είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η εξωτερική δράση, η ασφάλεια κτλ. Και επίση έχουμε 360 συγκεκριμένε δράσει Τίποτα το λιγότερο. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ε, εμφανίστηκε εδώ η κυρία Μάλστροκ, ε, Άστρομ και η κυρία Ρέντινγκ. Ε, εμείς τι θα κάνουμε, θα εγκρίνουμε απλώς το σχέδιο δράση με μια σειρά ερωτήσεων και με δύο κράσεις των επιτρόπων. Δηλαδή ούτε καν δεν θα τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, δεν θα έχουμε κάποιο ψήφισμα δεν θα κάνουμε κάτι. Έτσι λοιπόν εκφράζω εδώ την αντίρρησή μου ως προς τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που ακολουθείτε. Δεν μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε 360 συγκεκριμένες δράσεις ε, απλώς με κάποιες ερωτήσεις που θέτονται εδώ και με την ακρόαση Επιτρόπου και επίσης ε, να ρωτήσω την κυρία Μάλστρομ, την οποία φυσικά την ευχαριστώ για την παρουσία της εδώ. Η Ευρωπόλ 2013, γιατί θα έχουμε κανονισμό, δεν μας ε, φτάνει η απόφαση του Συμβουλίου. Δεύτερη ερώτηση μία πρόταση σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Ευρωπόλ, Eurojust και Frontex. 2011 ε, ε, είναι ο ορίζοντας. Και γιατί θα έχουμε μια σχετική πρόταση με την Ευρωπόλ και με το Situation Center, ε, δηλαδή ποιες είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Ευρωπόλ και το Situation Center. Επίση, οι νομοθετικέ προτάσει που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του Eurosur για το 2011, ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και γιατί ε, τελικά πρέπει να περιμένουμε στο 2014 για να κάνουμε αξιολόγηση τη οδηγία περί επιστροφών. Ευχαριστώ και γιατί πρέπει να περιμένουμε, όπω σα είπαμε, το 2014 για την αξιολόγηση αυτή τη οδηγία επιστροφών. Κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μάστρο. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το πρόγραμμα TFTP, το συζητήσαμε ήδη και με τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και αν η Ευρώπη δεν έχει αυτούς τους απαραίτητους μηχανισμούς, ε, ποια πρωτοβουλία θα έπρεπε να θα μπορούσε να αναλάβει η Κομισιόν προς την κατεύθυνση αυτή, αν και ξέρουμε ότι εδώ μιλάμε για πρωτοβουλία των τρίτων μελών για τη μετανάστευση, τι θα γίνει με την ε, κοινή μεταναστευτική πολιτική και με την κοινή πολιτική ασύλου, θα περιοριστούμε στις ε, κοινέ πτήσεις ε, επιστροφής, επαναπατρισμού και επίσης στη συνεργασία με τρίτες χώρες και στις συμφωνίες επενδυτοχής. Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά το πακέτο για τη βία Ε, πραγματικά να σας πω ότι αν συνεχίσετε ε, να εργαστείτε επί του θέματος ε, της ε, σεξουαλικής κατοικοποίησης και της εμπορίας ανθρώπων, είστε ξέπαινοι αλλά για την ε, ε, βία κατά των γυναικών ε, θα συνεχίσετε να εργάζεστε. Πιστεύετε ότι οι αριθμοί που δίνουν σήμερα κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η WAY, η οποία έχει έδρα στην Αυστρία, για 11.500 ε, γυναίκες στην Ευρώπη οι οποίες δολοφονούνται ε, λόγω αυτού του φαινομένου της βίας που ασκείται εναντίον τους. Ε, είναι απίστευτος ο αριθμός αυτός, επομένως τι θα κάνει η Κομισιόν θα θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και πώς μπορούμε να προλάβουμε τη βία αυτή. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπάουρ. Thank you so much for this opportunity and allow me to follow. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και θα ήθελα να ακολουθήσω την ευθεία γραμμή της συναδέλφου ρωτώντας σας ποιο θα είναι το μέλλον για την προτάσεις της Ισπανικής Προεδρίας αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την βία κατά των γυναικών. Όπως γνωρίζουμε από την εμπειρία της Ισπανίας, είναι περισσότερο δικαστικό ζήτημα παρά στατιστικής φύσης. Γι' αυτό θίγω το ζήτημα τώρα και εδώ, διότι θα πρέπει να το δούμε το ζήτημα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα τώρα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την ε, σωματεμπορία και την εμπορία ανθρώπων. Άκουσα την πρότασή σας, υπάρχουν όμως κάποια κρυμή ζητήματα γιατί έχει ελαττωθεί το μέγιστο της ελαχής της ποινής από 6 σε 5 και από 12 σε 10 έτη. Σε ό,τι φορά την ε, προστασία των θυμάτων, Ουσιαστικά η πρόταση ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, π.χ. στις περιπτώσεις ε, πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά και όχι στην επαγγελματική κατάρταση. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε και κάποιες πληροφορίες ανησυχητικέ που προέρχονται από το Συμβούλιο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και πώς πρόκειται να εξελιχθούν. Σας ευχαριστώ. Θα διαπιστώσατε πως δέθησαν διάφορες ερωτήσεις αναφορικά με τις, για θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της κυρίας Ρέντινγκ και όχι της κυρίας Μάλστρομ για θέματα θεμελιδών δικαιωμάτων και δικαιοσύνης. Το υπενθυμίζω λοιπόν αυτό και παρακαλώ να εστιάσουμε στα όσα μας είπε η κυρία Μάρτσον και στις αρμοδιότητές της. Ο κύριος Μασίπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι έχετε διάφορες δυσκολίες, όχι με το Κοινοβούλιο, αλλά με το Συμβούλιο. Πολύ δύσκολη λοιπόν για να προωθήσετε το ζήτημα του ασύλου αλλά και την πολιτική επανεγκατάσταση. Και μας ζητάτε ιδέες ε, ευρηματικές και μα ζητάτε την συνεργασία μας. Μα τη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη μας την έχετε. Την χάνετε της εμπιστοσύνη μας και όλα αυτά καταδεικνύονται απόλυτα με το όνομα της Επιτροπής. Ελευθερίε, πολιτικές ελευθερίες. Εσείς είστε υπέρμαχο των πολιτικών ελευθεριών και εγώ το ίδιο μου ότι δεν ανήκω στον δικό σας πολιτικό χώρο. Ε, σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και το τονίζω. Τώρα σε ό,τι φορά τις ε, δημιουργικές και ευρηματικές ιδέες έχω στο μυαλό μου μία, δηλαδή να εντοπίζουμε τα προβλήματα που αφορά στην πολιτική ασύλου και πρέπει λοιπόν να τα εντοπίσουμε σε υπόψη τι ε, κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχουν σε όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο για το ζήτημα των προσφύγων, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν μιλάμε μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για όλα τα άλλα, τα κοινωνικά κλπ. Και τέλος να σας πω ότι όπως εγώ σας στηρίζω και σα εκφράζει την εμπιστοσύνη μου, θα ήθελα να πω ότι μου ενέπνευσε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη την ε, Ολομέλεια προχθές ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν με τις ιδέες του και με τα όσα μας είπε και τα όσα άκουσα και από τους συναδέλφους που επισκέφθηκαν προσφάτως στην Ουάσιγκτον. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας ιστορικής συμφωνίας και θα πρέπει και από τις δύο πλευρές της Ατλαντικού να πετύχουμε μια μεγάλη και σημαντική συμφωνία πάνω σε θέματα ελευθεριών όπως τα εξέφρασε πολύ ορθά ο Αντιπρόεδρος Μπάιντεν. Οι δισταγμοί λοιπόν θα πρέπει να ξεπεραστούν. Και για μια ακόμα φορά τονίζω ότι έχουμε απόλυτη του πρόσωπό σα. Κύριε Φατζόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε για τις πληροφορίε. Έχω μια ερώτηση σχετικά με το σύστημα Schengen Δεύτερη γενιά. Είπατε ότι περιμένετε την ακριβή υπολογισμό για την περαιτέρω χρηματοδότηση. Υπολογίζω ότι θα υπάρξουν περαιτέρω έξοδα και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τη χρηματοδότηση αυτού του συστήματος. Αν το, και αν το κόστος ε, θα είναι υψηλότερο, πόσο υψηλότερο πιστεύετε ότι θα είναι. Και η άλλη ερώτηση που έχω να σας θέσω αφορά το ΣΥΣ 2. Πόσο θα διαρκέσει φυσικά και πόσο θα αυτή η καθυστέρηση η οποία προβλέπετε θα μας οδηγήσει το συντισμό δυνατόν στο να βρούμε ένα σύστημα το θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Τώρα, για τις ε, προξενικές θεωρήσεις, μία από τις προτεραιότητες που αναφέρατε και πάνω σε αυτό έχουμε ανταλλάξει πανδηλημένα γνώμες ε, στις συζητήσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Ποσνία, Ριζογοβίνη και την Αλμπανία. Είπατε ότι ελπίζετε πως ε, σύντομα θα προτείνεται την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω από τι ακριβώς εξαρτάται. Άκουσα κάποιες θετικέ ε, αξιολογήσεις, ε, ότι παραμένουν κάποια θέματα ακόμα ανοιχτά για κάποια κράτη, αλλά ε, Άκουσα επίσης ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, ασχολείστε και τον, επιμένετε επί των τεχνικών κριτηρίων μόνο ή η πολιτική κατάσταση θα μπορέσει μάλλον να επικρατήσει. Ξέρουμε ότι στην Αλβανία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά πιστεύω πως και οι δύο χώρες έχουν το σύντομο ανάγκη από τον Τουσταλή ένα θετικό μήνυμα του σύντομων δυνατών σε ρωτώ λοιπόν, περιμένετε να πέσει αυτή η απελευθέρωση μέχρι τα τέλη του έτους και προτίθεστε να στείλετε άμεσα τους εμπειρογνώμονές σας κάτι που δήλωσε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη είπε ότι θα μπορούσαν να φτάσουν ήδη αύριο. Εσείς πόσο καιρό νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Λέντ. Να σας πω ότι δεν ε, έριξα μια ματιά στο σημείωμα της συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ σχετικά με το συζητήριο, διότι ήμουν σκιώδης θηγητής για το σύστημα αυτό. Την προσεχή εβδομάδα στο Στρασβούργο οι εκθέσεις αυτές ε, θα περάσουν προψήφιση από την Ολομέλεια και εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών οι δύο αυτές εκθέσεις ψηφίστηκαν και έγιναν δεκτές κάποιες τροπολογίες οι οποίες εξέφεραν τις ανησυχίες μας αναφορικά με το κόστος και την ιδιαίτερη καθυστέρηση που παρουσιάζουν τα δύο αυτά προγράμματα. Ε, και κάτι άλλο. Μας ανησύχησε ιδιαίτερα η έλλειψη διαφάνειας ε, απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΣΥΣ αποτέλεσε επιτυχία και θα θέλαμε το ίδιο να συμβεί και με το συς Και οι φήμες ε, που φτάνουν στα αυτιά μας ε, δεν ε, μας διασκεδάζουν τις ανησυχίες μας, ιδιαίτερα κάποιες φήμες από πλευράς Συμβουλίου. Έως εκ τούτου ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει τυπικά σχετικά με τα αποτελέσματα της τελευταίας δοκιμής που έγινε στο ΣΥΣ2. Για μια δεύτερη ερώτηση πιο σύντομη, σχετικά με την συζήτηση η οποία έγινε αναφορικά με τους ε, εργαζομένους τρίτων χωρών που φτάνουν στις ε, αγορές εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω κατά νου τους, ε, επίσης και τους εργαζομένους που προέρχονται από, νέα, από τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε να δουλέψουν στις, στα παλιά κράτη-μέλη. Θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη τα οποία διατερούν περιορισμούς για τους εργαζόμενους που προέρχονται από τα ε, ενταχθήσεις ε, χώρες ε, να άρουν αυτούς τους περιορισμούς. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγιγιών, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ασχοληθώ με το ζήτημα του ασύλου. Είπατε ότι τα κείμενα είναι περίπλοκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ε, δυσκολίες κλπ. Το κατανοούμε. φυσικά θα θέλαμε να δεχτείτε τις ιδέες μας αναφορικά με την άρση αυτών των εμποδίων. Αλλά στο πρόγραμμα δράσης δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη λήψη μέτρων για την άρση των, των εμποδίων. Επιτρέψτε μου να σας ε, επαναλάβω για μια ακόμη φορά την ερώτηση πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αλληλοβοηθούμε για να άρουμε τα εμπόδια. Και το... Τώρα μια δεύτερη ερώτηση που θα θέλω να υποβάλω αφορά τους ε, μετανάστες ε, και την αγορά εργασία. Στο κείμενο που μα παρουσιάσατε, άκουσα κάποιε αναφορέ άμεσε αναφορικά με την πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασία. Στην γαλλική εκδοχή διαβάζω μια συντονισμένη πολιτική σύμφωνα με τι ανάγκε τη εθνική αγορά εργασία. Νομίζω ότι και σε άλλε γλώσσε το αυτό θα λέγεται. Και να σα. Δεν θα ήθελα να σα δώσω κάποια παραδείγματα, αλλά θα ήθελα να μα διαφωτίσετε σε αυτή την ε, πτυχή που αναφέρεται στο κείμενο και που ο μετανάστες θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις δημογραφικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κάποιες ε, δηλώσεις να μας κάνει τώρα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Το κείμενό σας τονίζεται την αυξημένη προστασία. Ένα από τα κράτη-μέλη ε, προωθεί ένα κείμενο της ε, συμφωνίας που έχει με τη Ρουμανία για επιστροφή των συνοδεύτων ανηλίκων που παρομοιάζει με απέλαση των ε, ασυνοδεύτων ε, ανηλίκων. Και θα ήθελα να γνωρίζω εάν έχετε την εντύπωση ότι η λόγω χώρα μέλος ε, πραγματικά εφαρμόζει αυτή την επιλογή που επιλέξατε κι εσείς για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κύριε Παδοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, όντω θεωρώ ότι είναι πολύ φιλοδοξία η ατζέντα σα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σα ότι χρειάζεται πολιτική εναρμόνιση των πολιτικών στι πολιτικέ ασύλου και ενίσχυση τη κοινωνικής αλληλεγγύη, ιδιαίτερα προ τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου που μαστίζονται από την νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Το ερώτημα μου είναι σαφές ένα σχέδιο δράση πρέπει να έχει σαν στόχο να μετατρέψει στόχου και προτεραιότητε του προγράμματο τη Στοκχόλμη σε συγκεκριμένε δράσει με σαφέ χρονοδιάγραμμα υιοθέτηση και εφαρμογή. Θεωρώ ότι τα θέματα ασύλου, μετανάστευση και μη διάκριση δεν είναι καθόλου ενισχυμένα μέσα στο σχέδιο δράση. Χρειάζεται να υπάρχει επιτάχυση και μηχανισμοί υλοποίηση, όχι να μένουμε απλά σε θεωρίε. Και το ερώτημα μου είναι πώς μπορεί να κινηθούμε με πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί μέχρι ότου βρούμε χρυσές τομές, η λαθρομετανάστευση μαστίζει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Το δεύτερο ερώτημα αναφορά το πιλωτικό πρόγραμμα που γίνεται στη Μάλτα. Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για να έχουμε αυτά αποτελέσματα, και να δούμε πώς προχωρούμε. Και το τρίτον, έχετε εκφράσει ικανοποίηση για την πρόοδο όσον αφορά τη Συμφωνία Επανεγκατάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Γνωρίζω ότι αυτή η συμφωνία εκκρεμεί από το 2002. Βρισκόμαστε στο 2010. Πότε θα είστε σε θέση να παρουσιάσετε ολοκληρωμένη αυτή τη συμφωνία και να μπει σε εφαρμογή. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Όταν στη σελίδα 3 αναφέρεστε ότι η Κομισιόν θα επιδιώξει να επιδείξει μηδενική ανοχή σε παραβιάσεις στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τι θα κάνει δηλαδή έμπραχτα σε χώρες που παραβιάζουν τα δικαιώματα, παραδείγματο χάρη είτε των μεταναστών, είτε το Ρώμα, είτε ανθρώπινα δικαιώματα. Έμπραχτα. Thank you. Thank you. Colleagues. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει και Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών, αλλά αν σεβαστείτε το χρόνο, ένα λεπτό ο καθένας, να σας δώσουμε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε. Κυρία Ματιά, ευχαριστώ. Θέλω να θέσω μια ερώτηση στην κυρία Μάλστρομ ε, γιατί η απαντήση που έδωσε στους συναδέλφους ε, σε ό,τι αφορά τους ε, εποχικούς εργαζομένους δεν με έπεισε. Θα ήθελα να μου πείτε πότε ακριβώς σκοπεύετε να παρουσιάσετε την πρότασή σας για αυτούς τους εποχικούς εργαζομένους γιατί έχουμε την εντύπωση ότι καθυστερεί. Και η απάντηση που δώσατε δεν με έπεισε. Θέλω συγκεκριμένη ημερομηνία σας παρακαλώ κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ. Κυρία Μακοβή, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Μάλστρομ για την παρουσία τη. Ε, Όπω ξέρετε, την περσμένη εβδομάδα υιοθετήσαμε μια γραπτή δήλωση κατά τη διαφθορά που ζητά από την Κομισιόν να συστήσει ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση της διαφθοράς στα κράτη-μέλη. Πώς ε, σκοπεύετε να απαντήσετε σε αυτή την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ανάληψη δράση στον τομέα αυτό, κύριε Μπρόντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του συστήματος θεωρήσεων, θέλω να θέσω μια ερώτηση στην κυρία Μάλστρομ. Ε, την περσμένη εβδομάδα έγινε μια συζήτηση και προσεγγίσαμε διάφορα ζητήματα. Κυρίως αναφερθήκαμε στη Βοσνία. Το Σύνταγμα της Βοσνίας αποκλεί τους Εβραίους από το να λάβουν κάποιες ε, υψηλές διοικητικές θέσεις επιπρόσθετα ε, οι θρησκευτικοί ηγέτες ε, ήθελαν να συμπεριλάβουν και τις σειρά στο Σύνταγμα. Υπήρξε και μία ε, σε ένα χωριό στην Βοσνία κάποιοι πήραν τα όπλα και είχε εισαχθεί η Σαριά και μάλιστα να σας πω ότι βλέπουμε και κάποια τρομοκρατική δράση στη Βοσνία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Είστε ε, ενήμεροι επίσης στην Αλβανία. Έχουμε και ε, κάποιες επιθέσεις κατά των ομοφιλοφίλων. Τα γνωρίζετε όλα αυτά τα συμβάντα, όλα αυτά τα γεγονότα σε αυτές τις δύο χώρες. Και μια ακόμη ερώτηση όταν πρόκειται και το άσυλο και για τη μετανάστευση. Ελπίζω ότι το πακέτο αυτό ε, δεν θα ψηφιστεί. Ήδη η χώρα μου έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με την ένταξη κατόπιν μαζικής μετανάστευσης. Εμείς θέλουμε μία μη κεντροποιημένη, μη κεντρική πολιτική. Θέλουμε μια πολιτική που θα καθορίζεται από την ίδια τη χώρα, από το ίδιο κράτος μέλος. Ποια θα είναι η δική σας στάση όταν μια χώρα θέλει να χρησιμοποιήσει το προηγούμενο καθεστώς όπως έκανε η Δανία παραδείγματος χάρη και δεν επιθυμεί να εφαρμόσει ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλετε το λόγο, ε, γιατί έχουμε καθυστερήσει και νομίζω ότι μάλλον θα δυσκολευτεί να απαντήσει και η κυρία Μάλστρομ. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να κάνετε λιγότερο από ένα λεπτό. Να δώσουμε σε εσάς το λόγο. Ευχαριστώ. Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Μία απλή ερώτηση. Στα πλαίσια του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους ε, πρόσφυγες, θα υπάρξει πρωτοβουλία από την Επιτροπή για την ανάπτυξη και δημιουργία προγράμματος εσωτερικής επανεγκατάστασης για τους πρόσφυγες. Το συζητήσαμε στα πλαίσια του resettlement. Ε, δεν έχουμε όμως συγκεκριμένο προγραμματισμό από την Επιτροπή. Και στα πλαίσια της ε, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, το θεωρούμε σοβαρή προτεραιότητα και θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση. Thank you. Ευχαριστώ. Θα δυσκολευτεί μάλλον κυρία Μαστρόμ να απαντήσει σε τόσο πολλέ ερωτήσει, αλλά φανταζόμαι ότι θα μπορέσετε να δώσετε κάποιε συλλογικέ απαντήσει στα όλα ακούστηκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω το πρόγραμμα δάση στο Κόλμης αποτελεί ένα κατάλογο προτάσεων και προσπαθήσαμε να λαβούμε υπόψη και θέματα που απασχολούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρονται στο σχετικό ψήφισμα. Φυσικό είναι πολύ αποτελεσματική η Κομισιόν. Κάποια θέματα θα σας παρουσιαστούν ε, ακόμη και πριν την υλοποίηση του προγράμματο δράση τη Και φυσικά δεν αποκλείω ότι θα προκύψουν και άλλα. Βέβαια, έχουμε και ορισμένα εκκρεμή θέματα από την προηγούμενη Κομισιόν και όπω είπε και ο Πρόεδρο, κάποιε από τι ερωτήσει σα ό,τι αφορά ε, την βία κατά των γυναικών, ε, ένα θέμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι τομέα τη κυρία Ρέντινγκ αυτό. Έτσι λοιπόν, θα τη ζητήσω όταν θα έρθει εδώ να σα επισκεφθεί, να αναφερθεί αναλυτικά στο ζήτημα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την αλληλεγγύη, ο κ. Ζικολίνο έθεσε μια ερώτηση. Νομίζω ότι πολλά ήδη έχουν γίνει για την αλληλεγγύη. Η Κομισιόν προτείνει ένα θεωρημένο μηχανισμό του Δουβλίνου προκειμένου να λάβει υπόψη την έντονη πίεση που ασκείται προσωρινά σε ορισμένα κράτη-μέλη. Κάποια μέλη το έχουν ζητήσει τώρα εξολογούμε το πρόγραμμα της Μάλτας και έχουμε μεταφορά ορισμένων ανθρώπων στα πλαίσια του προγράμματος αυτού από τη Μάλτα θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε να έχουμε ένα πιο μόνιμο μηχανισμό. Τώρα ε, σκορπεύουμε να ανακοινώσουμε και μια πρόταση για την ενισχυμένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φαντάζομαι ότι θα δοθούν και άλλα κίνητρα προκειμένου να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη. Κύριε Λαμπρινίδη για την Τουρκία. Ναι, Όλοι, όλοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία επενδυτοχή. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία τώρα, αλλά είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ξέρω ότι κράτησαν πάρα πολύ, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες ε, σημειώσαμε πρόοδο και ε, πραγματικά ευχαρίστω να σα δώσω στο μέλλον περισσότερε λεπτομέρειε. αλλά είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τη διαδικασία για το SWIFT. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε και συζητούμε με του Αμερικανού. θα δούμε που θα καταλήξουμε για την ένταξη. Ναι, η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει στην Κομισιόν νέε αρμοδιότητε. σχετικά. Έχουμε μόλι εκδώσει το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο με παραδείγματα από όλα τα κράτη-μέλη, γιατί φυσικά η ένταξη γίνεται καλύτερα σε τοπικό επίπεδο, του χρόνου η Κομισιόν θα παρουσιάσει ένα σύνολο κριτηρίων και μεθόδων που μπορούν να συνδράμουν στην καλύτερη ένταξη και φυσικά θα ανταλλάξουμε και πάρα πολλές διασκέψεις για την ε, διαφθορά, κύριε Ράτφορντ. Μάλιστα, είστε. Κι άλλο συναδελφό σα το ρώτησε, ναι, θα παρουσιάσουμε μέχρι το τέλο του έτου μια ανακοίνωση για τη διαφθορά και θα δούμε πώ μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό αξιολόγηση για το θέμα αυτό. Για τη διαφθορά στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μα εναντί και άλλων χωρών που υποστηρίζουν την καλή διακυβέρνηση και την δημοκρατία. Πρέπει και σε ιστορικό επίπεδο να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. για τους συνεροφυλάκες της Frontex. Ε, ναι, ζητήθηκε από την Κομισιόν να το ξελογίσει το θέμα αυτό, δεν είναι πρόταση. Για την εξωτερική διάσταση του ασύλου και τη ε, περιφερειακή συνεργασία να συνεργαζόμαστε με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξη. Συζητώ συχνά με τον κύριο Πίμπαλξ και νομίζω ότι θα αξίδει η συνεργασία μα ε, στο μέλλον για τις ιστοσελίδες ε, παιδικής πορνογραφίας. Ε, έχουμε ε, μεγάλη τεκμηρίωση και από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και από τις ΜΚΑΠΑ Όμικρον. Ευχαρίστω να σας δώσω ορισμένες διευθύνσεις που μπορείτε να τις ελέγξετε κι εσείς. Καταπολεμής της τρομοκρατίας, κυρία Ρομέρο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό κάνουμε μία αξιολόγηση όλων των μέσων και των μεθόδων που έχουμε ήδη στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε αν υπάρχει κάτι που λείπει, αν υπάρχει ένα κενό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα σε ό,τι αφορά την πρόληψη για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερες, ό,τι φορά το συντονισμό, την προστασία των υποδομών και την προστασία των θυμάτων. Και θα προτείνουμε πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Στις δύο. Ναι. Βεβαίως είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό που το κληρονομήσαμε. Ίσως ε, να μην είναι και ένα από τα καλύτερα δώρα που μας έδωσε η προηγούμενη Κομισιόν. Ακολουθήσαμε τον ε, οδικό χαρτί του Συμβουλίου κατά γράμμα, προσπαθήσαμε να είμαστε στον το πιο και εγώ προσπαθήσα να το δω με μια νεμετιά τώρα. Το πρώτο μάλιστον, ε, η πρώτη δοκιμή μάλιστον ήταν επιτυχής και φυσικά οι εμπειρογνώμες των κρατών μελών συμμετέχουν στην αξιολόγηση τώρα θέλουμε να δούμε ποια θα είναι τα μελλοντικά βήματα, ο προπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα που θα μα οδηγήσουν στο δεύτερο μάλιστον, το φθινόπωρο. Και ελπίζω να τα παρουσιάσω όλα αυτά σύντομα τον Ιούλιο ή αμέσω μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Έχω γράψει και μια επιστολή στον Πρόεδρο και στον κύριο Κοέλιο για να τον ενημερώσω σχετικά Ελπίζω να έχει διανεμηθεί η επιστολή αυτή στην Επιτροπή και θα συνεχίσω φυσικά να παρέχω όσο δυνατόν περισσότερο διαφανεί πληροφορίε, γιατί ξέρω ότι σα ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Και δεν θέλω τώρα να κάνω μία εκτίμηση του τελικού κόστους, αλλά φυσικά ε, θα πρέπει να μας αποπληρώσουν ε, και ένα ποσό η αναδοχή λόγω των καθυστερήσεων. γιατί η Βοσνία Ερζεγοβίνη συνεργαζόμαστε με τη χώρα αυτή σε τεχνική βάση, γιατί είναι αντικειμενικά και διαφανή τα κριτήρια και οι δύο χώρες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Ε, συνεργαζόμαστε τώρα μαζί τους και σε επίπεδο πυρογνωμόνων κρατών μελών για να δούμε πόσο θα χρειαστεί, πόσο χρόνο θα χρειαστεί ακόμη για τις χώρες αυτές. Ε, δηλαδή να δούμε αν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα ή αν θα μπορούμε να πούμε ένα ναι, υπό πόρους. Σε κάποιες εβδομάδες θα το γνωρίζουμε. Σε ό,τι αφορά την νόμιμη μετανάστευση πριν από το καλοκαίρι, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα την παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή. Θα έλθει η πρόταση πριν το καλοκαίρι. Η Κομισιόν έχει τόσε πολλέ προτάσει. Ε, έτσι λοιπόν, είμαστε σε διαπραγματεύσει με το Γενικό Γραμματέα για να δούμε ποια θα είναι ακριβή ημερομηνία που μπορώ να την παρουσιάσω στο Σώμα των Επιτρόπων. Αλλά πριν το καλοκαίρι σα το υπόσχομαι. Δεν ε, υπάρχει εδώ πολιτική... μια πολιτική σκοπιά που θα πρέπει να εξετάσουμε για του ασυνόδευτους ανηλίκους. Ναι, μία από τις προτάσεις είναι ότι κάθε παιδί θα πρέπει να έχει έναν ε, ε, νομικό εκπρόσωπο που θα το παρακολουθεί σε όλη τη διαδικασία. Ελπίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα δεκτούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφθορά, μάλιστα. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Προσπάθησα, τουλάχιστον. Έβαλα δυνατά μου ορισμένα από τα θέματα, τα οποία αναφέρθηκαν ε, εντάσσοντας τις αρμοδιότητες κυρίας Βέντινγκ. Φαντάζομαι ότι θα έλθει και αυτή στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλστρομ ε, μας ε, απάντησε. και πραγματικά εκτιμούμε τις προσπάθειές σας να συνοψίσετε στις απαντήσεις σας, ε, όλα τα θέματα που τέθηκαν και φυσικά βλέπουμε ότι αυτές τις συναντήσεις πρέπει να τις υλοποιούμε όσο το δυνατόν πιο συχνά. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Είδαμε πόσες πολλέ ερωτήσει τέθηκαν και φυσικά θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα σας καλούμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε να έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί βλέπετε ότι έχουμε ερωτήσει και απαντήσει να ανταλλάξουμε. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ, θα προσοχή. περάσουμε τώρα στο σημείο 4. Διαδικαστικό κύριος Κλέης. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Πάει καιρός ε, που είχε προσκληθεί η κυρία Επίτροπο στην Επιτροπή μας και κάθε φορά διαπιστώνουμε πως ε, όταν έρχεται ανάμεσά μας ε, γίνονται πάρα πολλές ερωτήσεις και γι' αυτό όπως είπατε, χρειάζεται να την προσκαλούμε συχνότερα ή να αφιερώνουμε και περισσότερο χρόνο. Με μια μισή ώρα που προβλεπόταν για σήμερα πάνω από τα... Οι συνάδελφοι δεν είχαν ε, αρκετό χρόνο για να μιλήσουν. Χρειάστηκε λοιπόν να κάνουν σύντομες παρεμβάσεις. Άρα προσκαλούμε συχνότερα. Εντάξει, θα συμφωνείτε πως ε, είναι γεγονός, ε, το σημειώνουμε, υπολήθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις και θα πρέπει να επισπεύσουμε λοιπόν τις επαφές μας με την ε, κυρία Μάλστρομ και να τη ζητήσουμε να έρχεται ως τιμό των δυνατόν στην Επιτροπή μας διότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά όπως βλέπετε ξεπεράσαμε κατά πολύ τον χρόνο ομιλίας, μάλλον τον χρόνο της ε, συνάντησης με την κυρία Επίτροπο και ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να απαντήσει στις περισσότερες των ερωτήσεων. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4 της μισής διατάξεως μέτρα επιτροπολογίας ε, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των θαλασσίων συνόρων Frontex Πρόκειται για ένα αίτημα της ε, Γιούρη σχετικά με την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό το ζήτημα αφορά την ε, απόφαση του Συμβουλίου για το Frontex. Ε, θα θυμίστε ότι επανειλημμένα συζητήσαμε την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τον κώδικα συνόρων και την εφαρμογή του σε περιπτώσει που η Frontex παρεμβαίνει στην θάλασσα. Η απόφαση του Συμβουλίου που πρόσφατα δημοσιεύθηκε θα θεωρήθηκε από την Euro ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στο δικαστήριο και θεώρησε ότι τα ζητήματα που θίγει η απόφαση θα έπρεπε να βασίζονται σε μια πιο σταθερή νομική βάση. Ένα σχέδιο επιστολή λοιπόν στην ε, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, συντάχθηκε και διενεμήθη σε όλους σας. Προτείνω λοιπόν να υποστηρίξουμε το κείμενο της επιστολής και διαπίστωσα ότι ο κύριος Μπουζουτήλ πρότεινε να ζητήσουμε από το δικαστήριο να υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης ε, μέχρι τη, αυτής της επιστολής μέχρι τη στιγμή που η πράξη θα εγκριθεί ολοκληρωτικά βασιζόμενη σε πιο σαφή και στεναρή νομική βάση. Ο κύριος Κάσμαν είδα ότι ζήτησε το λόγο, μετά κυρία Τζανίνου, κύριε Κάσμαν. Α, είδα που ένευε η Σανίν, ήθελα να με χαιρετήσει, χαιρετώ και εγώ. Λοιπόν, πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η ομάδα μου ψήφισε υπέρ του μέτρου όπως ξέρετε, αναγνωρίζοντας ότι η νομική βάση δεν ήταν η κατάλληλη. Αποφασίσαμε τα μέτρα όμως ότι ήταν ε, κατεπήγοντα και αναλογικά. Ερωτήσεις. Στην επιστολή και στην τελευταία παράγραφο σίγουρα επαναλαμβάνουμε ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθούν τα μέτρα αυτά μέχρι ότου το δικαστήριο ε, αποφανθεί τι διασφαλίσεις μπορείτε να μου δώσετε ότι το περιεχόμενο αυτό θα ληφθεί απόλυτα υπόψη από την Νομική Επιτροπή. Δεύτερον, δεδομένης της δέσμευσης του κυρίου Μπουσουτήλ και της δήλωσής του στο Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση, τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων πριν από την ψηφοφορία, ότι θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία. Ε, ο κύριος Μπουσουτήλ θα ε, ε, προσέθεται στην οδηγία Frontex τα μέτρα αυτά για να ε, γίνεται η έρευνα και η αναχέτηση που θεωρούμε ότι χρειάζεται επί τη βάση των απαντήσεων που θα λάβουμε, η ομάδα μου θα αποφασίσει τι στάση θα κρατήσει στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Η κυρία Χένις Πλάσερτε, είδα το χέρι σα. Όχι, όχι, δεν ζήτησα. Ε, εγώ ήθελα, ήθελα να κάνουμε ψηφοφορία κυρία Γκάνς. Και εγώ το ίδιο ήθελα να πω, όπως ο κύριος Κάσμαν. Το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό για μας και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα είναι ανασταλτικό αν ψηφίσουμε υπέρ της επιστολής. Δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα αν ψηφίσουμε υπέρ της επιστολής. Κυρία Βέμπερ. Το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η αρμοδιότητα κάθε θεσμικού οργάνου της Ένωσης. Αν υπάρχει υποψία ότι κάποιες εξουσίες έχουν υπερβαθεί, θα πρέπει το δικαστήριο να αποφανθεί αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Ε, οπότε η οχι οποτε η ομαδα μου θα ψηφίσει υπέρ. Διατυπώθηκαν ερωτήματα απευθεία στον κύριο Μπουσουτήλ. Σάιμον, ευχαριστώ αν κατάλαβα καλά. Δύο ερωτήσεις ακούσαμε. Η πρώτη είναι για την νομική υπηρεσία. Αν εκπροσωπείτε εδώ, ας απαντήσει, είναι δικό του θέμα. Τώρα, για την ερώτηση προ εμένα, αν προτίθεμε να συμπεριλάβω, να δεχτώ να συμπεριληφθούν στην πρόταση Frontex τα μέτρα αυτά για την οποία είμαι εισηγητής. Εγώ δεν είμαι ε, εκείνο που λαμβάνει την πρωτοβουλία για την ε, νομοθεσία. Εγώ είμαι εισηγητή του Κοινοβουλίου Κομισιόν. Θα το κάνει αυτό. Και έχουμε και πρόταση επιτάπητο. Είμαι ανοιχτό να συνεργαστώ με του κοιόδη εισηγητέ, να δούμε τι πιστεύουν και εκείνοι και να συμφωνήσουμε κάπου. Υπενθυμίζω όμω ότι παρά την ε, αναθεώρηση της εντολής του Frontex, που είναι η πρόταση που έχουμε εδώ, αυτά τα μέτρα είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι τώρα ήδη πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή ανεξάρτητα από την πρόταση για το, την πρόταση για το Frontex. Είναι δύο διαφορετικά θέματα μέχρι τώρα. Αν υπάρξει συμφωνία με τους σκιώδεις, ούτως ώστε να ληφθούν αυτά υπόψη και να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα νομική πτυχή, ίσως η νομική υπηρεσία του, του Κοινοβουλίου θα ήθελε να σχολιάσει. Όχι. Όχι. Α. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. νομική υπηρεσία. Πράγματι, ε, ε, το αίτημα για την διατήρηση της ε, πράξης σε ό,τι αφορά την απόφαση η οποία έχει προσβληθεί ε, γίνει δεκτή. Και, και τι γίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα, ας ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η πρόταση έγινε δεκτή. Ας προχωρήσουμε. Σημείο 6. Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον σχέδιο προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο τμήμα 3 Επιτροπή. Σκοπός είναι εδώ ανταλλαγή απόψεων. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον προπολογισμό του 2011. Αρχικά θα ακούσουμε την Κομισιόν και μετά τα μέλη που το επιθυμούν θα λάβουν το λόγο. Έχουμε προετοιμάσει ένα έγγραφο εργασίας Συγγνώμη, συγγνώμη, έκανα λάθος. Πρώτα έχουμε το σημείο 5 που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας. Έχουμε μια παρουσίαση σχετικά με την συνέχεια της ΑΣΟΚ και παρουσίαση κατάσταση των διαπραγματεύσεων του Συμβούλου. Από την τελευταία μας συνεδρία η κυρία Ματιό συνέχισε να εργάζεται επί αυτού του ευαίσθητου Ζητήματο, ε, συνάντησε την 5η Μαΐου το Ενκομισιόν και το Συμβούλιο για συζητήσει του σύμβασμού που είχαν εγκριθεί από τους σκιώδεις ε, Τώρα θα μας συνοψίσει σχετικά και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις 25 Μαρτίου η Επιτροπή Απασχόληση ψήφισε την ε, συμβολή της στο σχέδιο της οδηγίας. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο Πρώτα στην κυρία Ματιού, η συγκήτρια. Ακολούθησε τον κύριο Σέρκας. Αν παρευρίσκεται, δεν παρευρίσκεται. Ο συνεισηγητής από την Επιτροπή ΑΣΟΚ. Ας ακούσουμε όμως την κυρία Ματιού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, η Επιτροπή Απασχόλησης ε, ψήφισε το έγγραφό της ε, και την προηγούμενη εβδομάδα προχωρήσαμε σε έναν δεύτερο τριμερή διάλογο όπου καταλήξαμε σε κάποιες συμφωνίες ε, σχετικά με την Επιτροπή μας, την ΛΥΜΠΕ, σε θέματα τα οποία είμαστε αρμόδιοι στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας. Όλα βαίνουν πάνω κάτω καλώς, εκτός από ορισμένα σημεία τα οποία έχουμε κολλήσει, γι' αυτό το λόγο έλαβα και και τον λόγο κατά την παρουσία της κυρίας Μάλστρομ θα μας, θέλει να μας διευκρινίσει πότε θα προταθεί το σχέδιο της οδηγίας για τους εποχιακά εργαζόμενους διότι ακριβώς εκεί είναι που έχουμε κολλήσει και υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην Επιτροπή που έχει ήδη ψηφίσει αλλά και σε ορισμένες πολιτικές ομάδες προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εποχικά εργαζόμενοι στο πεδίο εφαρμογής. Στις 5 έχουμε μια συνεδρίαση με τους Κιώδης, άρα τώρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, διότι η ώρα είναι 5 παρα 10. Ποιες θα είναι η αντιδράση των πολιτικών ομάδων μετά από τη δηλώση της κυρίας Μάρστρομ, η οποία μας διευκρίνησε ότι θα υποβάλει την πρότασή της, μας το υποσχέθηκε πριν από τα τέλη Ιουνίου. Δεν ξέρω αν αυτό θα ικανοποιήσει όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο το οποίο έχει δυσκολέψει της, ε, την πρόοδο και έχουμε μια σειρά από συμβασμούς σχετικά με το θέμα αυτό της ε, ενίας άδεια, ε, κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να ξεκινάει αυτό το ζήτημα από το κράτος μέλος ή θα προέρχεται από το κράτος καταγωγής. Μπορεί λοιπόν αυτή η αίτηση να υποβληθεί από τον εργοδότη ή από τον ενδιαφερόμενο. Αυτά λοιπόν είναι σημεία των οποίων προσπαθούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Κατά τα υπόλοιπα δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα ανυπέρβλητα, αλλά ε, ούτε και αυτό που σας προανέφερα είναι ανυπέρβλητο. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε τάχιστα συμβαστικές λύσεις και τώρα την Ευήκον τις παρατηρήσεις σας. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας, εισηγητής από την Επιτροπή Απασχόλησης, δεν παρίσταται, αλλά ας ακούσουμε τον πρόσωπο της Κομισιόν και μετά τα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ. Πώς ονομάζεστε. Κυρία Όμεν, είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συνέντευξη. Χαίρομαι που σας βλέπω. Το όνομά μου δεν το έχω εδώ μπροστά μου, δεν έχω το καρτελάκι μου. Ίσως η γραμματεία να μπορούσε να με βοηθήσει. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Κύριε Πρόεδρε, είμαι η Σκιώδης Συγκίτρια. επί του θέματος ε, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και είχα την χαρά να ακούσω την κυρία Ματιό και χαίρομαι που δεν ε, βρίσκει να υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με τις που ενέκρινε η Επιτροπή μου. Ε, άρα λοιπόν τα εμπόδια όπως είπε δεν είναι υπέρβλητα. Ε, δεύτερον, ο λόγος που λαμβάνω το λόγο είναι ο εξής. Η κυρία Ματιό παρατήρησε πως υπάρχουν δυσκολίες ε, αναφορικά με το θέμα των εποχικά εργαζομένων. Αλλά αυτό το θέμα δεν το έχει εξετάσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά η δική σας. Και, Πρόεδρε, εάν ε, ήμουν μέλος της δικής Επιτροπής, ε, στην οδηγία αυτή δεν θα ήθελα να συμπεριληφθεί η εποχική εργασία, διότι ε, αυτή η εργασία είναι μικρής διάρκειας και πρόκειται για συνθήκες εργασίες που διαφέρουν σημαντικά όπως και το θέμα της κοινωνικής προστασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να την εξώσουμε με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Είναι ένα καθεστώς εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Να επαναλάβω λοιπόν πως στην Επιτροπή ΑΣΟΚ ε, δεν έχουμε συμπεριλάβει λοιπόν, το ζήτημα της εποχικής εργασίας και καλό θα ήταν να μην το συμπεριλάβετε ούτε και εσείς. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επειδή η Λίλια δεν ε, παρίσταται, θα ήθελα να ήθελα να σας αναφέρω ποια είναι η θέση μας Ρωτήσαμε την κυρία Μάρστρομ για το θέμα των εποχικά εργαζομένων διότι εδώ ε, εμπίπτει το θέμα της, ε, των ίσων ευκαιριών. Σε ό,τι αφορά τον άτυπο τριμηρή διάλογο, υποστηρίζουμε τον ε, εισηγητή. Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μας ως ομάδα. Αφενός, η ανάγκη ύπαρξης ε, περαιτέρω εγγράφων, ε, διότι θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι σημαντικό. Και το άλλο ερώτημα είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει το κράτο μέλο για το ζήτημα τη ενή διαδικασία υποβολή αίτηση για τη χορήγηση άδεια διαμονή, ε, θα πρέπει αυτή η αίτηση. Μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή είτε να απορριφθεί σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία θα υιοθετηθούν αλλά στο πλαίσιο της απαραίτητης διαφάνειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουζουτήλ, ευχαριστώ. Σύντομα. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την θέση των σοσιαλιστών για τους εποχικά εργαζόμενους, αλλά ε, υποστηρίζω και την άποψη της κυρίας ε, Όμεν Ρόιτεν, ότι δηλαδή δεν είναι εδώ κατάλληλος χώρος για να εξετάσουμε το θέμα ακριβώς, λοιπόν, για αυτό το ζήτημα. Επανειλημμένα ζήτησα από την κυρία Μάλστρομ λίγου να μας καταστήσει σαφές ότι θα υποβάλει πρόταση σχετικά με τους εποχικά εργαζόμενους προκειμένου το ζήτημα αυτό να μην ε, παραμεληθεί. Και ανέφερε ότι θα φτάσει μια πρόταση εντός των προσεχών εβδομάδων για τους εποχικά εργαζόμενους. Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διαφωνία πάνω στο θέμα, διότι δεν εμπίπτει στο πλαίσιο αυτής της προτάσεως και θα και τα πράγματα εάν τις συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Εκτό μικρόφωνο, πρόεδρος, η κυρία Έλμστ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι φαίνεται από τις τροπολογίες ότι είναι καυτό το θέμα. Και δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Πού είναι τα κύρια προβλήματα που αναδείξαμε και στις διαβουλεύσεις. Καταρχήν το πεδίο εφαρμογής. Ήδη έχουμε πει πολλά και πολλά δεν έχουν ληφθεί υπόψη το θέμα δυσκολεύεται γιατί έχουμε διάφορες κατηγορίες μεταναστών εργαζομένων που έχουν διαφορετικά δικαιώματα ή δεν έχουν κάποιες κατηγορίες και είναι προβληματικό αυτό. Ωραία ακούγεται αυτή η ρύθμιση, αλλά βλέπουμε ότι έχει κενά και είναι και γραφειοκρατική. Επίσης, να δούμε ποιος θα υποβάλει την αίτηση, ποιος πρέπει να την υποβάλει. Για να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αν ο εργοδότης θα είναι εκείνο που θα μπορεί ή θα έπρεπε να κάνει την αίτηση. Αυτό θα σήμαινε ότι ο εργοδότης θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, θα πρέπει να καταπιαστεί και να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και βεβαίως θα μπορεί να ασκεί κάποια πίεση στον εργαζόμενο. Και αυτό είναι πρόβλημα για τον υποπρόσληψη εργαζόμενο. Ήδη από αυτό το λόγο θα είναι δύσκολο να απασχοληθεί εκεί και θα είναι και προβληματική η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σας θυμίσω... Ελπίζομαι ότι οι ρυθμίσεις σε περίπτωση ανεργίας ε, θα είναι αποτελεσματικές. Υπάρχει μια πρόταση, βέβαια το Συμβούλιο το βλέπει τελείως διαφορετικά το θέμα. Ελπίζω ότι ε, αν υπάρξει ανεργία θα υπάρχει και η δυνατότητα να μπορεί κανείς ε, να προσληφθεί αλλού ή εν πάση περιπτώσει να μην χρειαστεί να φύγει αμέσω από τη χώρα. Αυτή η σύνδεση δηλαδή εργασία, άδεια είναι σημαντικό θέμα. Και τέλος η παλιά αιτιολογική σκέψη 19 από την πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικό αυτό, το έχουμε πει. Δεν ξέρω, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με το αν θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή πρόταση. Άλλα σχόλια, άλλα μέλη. Το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα μας πει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Απλώς να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ματιά. Έχουμε εργαστεί πολύ οργανωμένα και επικοδομητικά μέχρι σήμερα. Η κυρία Ματιά εντόπισε τα κρεμή ζητήματα και πιστεύουμε ότι τα θέματα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν επαρκή λόγο για να μας εμποδίσουν να φτάσουμε στη συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε που ψηφίστηκαν από την Επιτροπή Επασχόληση, γνωρίζουμε ακριβώ ποια είναι τα θεμελιώδη θέματα για την Επιτροπή αυτή, ποια είναι τα πιο σημαντικά και θα ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει με το ίδιο επικοδομητικό πνεύμα, προκειμένου να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό ήθελα να πω έξω με τους Πρόεδρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράνιας. Έτσι λοιπόν κλείνουμε τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης. Υπερθμόν 6. Τώρα, ναι. Απόφαση του Κοινοβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο 3 3, Επιτροπή. Εδώ έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τον προπολογισμό του 2011. Θα ακούσουμε μια σύντομη παρουσίαση από την Κομισιόν και κατόπιν θα ανοίξουμε το λόγο, θα δώσουμε το λόγο για τη συζήτηση. 2011 θα είναι ο πρώτο ετήσιο προπολογισμών υπό τι νέε διαδικασίε τη συνδίκη Λισαβόνα. Έχουμε μια ανάγνωση στο Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Και αυτό σημαίνει ότι στην Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με την Επιτροπή Προπολογισμών πιο στενά από ό,τι στο παρελθόν, έτσι, ε, η Κομισιόν παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού 27 Απριλίου του 2010. Τώρα η Επιτροπή Προπολογισμού προετοιμάζει ένα σχέδιο έκθεση για το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν, εντολή για το τρεμερή διάλογο. Η συγγήτρια είναι η κυρία Τσε... Τσεβέσκα. Πολύ δύσκολο να το προφέρω το όνομά σας, συγγνώμη προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να αντιδράσουν σε αυτό το προηγούμενο δύο και να καταθέσουν ε, τροπολογίε για την έκθεση αυτή, κατευθείαν στην Επιτροπή Προπολογισμού, να έχουμε αυτή την πρώτη ενταλλαγή απόψεων σήμερα. Τα έγγραφα αναφορά, δηλαδή το σχέδιο προπολογισμού τη Κομισιόν, ένα έγγραφο εργασία ε, που συνέταξα εγώ. Αφορά την, την πρόβλεψη για το 2011 και έχουμε και όσο γράφει αναφορά σε ένα αντίγραφο της έκθεσης ε, της κυρίας Τετσερδέσκα που στέλνει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την περασμένη Παρασκευή. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Τετάρτη 12 Μαΐου το μεσημέρι στις 12. Τώρα να δώσουμε τον λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο κύριος Ντεμπράουερ. Είστε εδώ, μάλιστα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εσείς ε, κάνατε μια σύντομη παρουσίαση και νομίζω ότι αυτή την προχωρημένη ώρα πρέπει να είμαστε σύντομοι καθώς είχαμε ήδη την ευκαιρία να δώσουμε στην Επιτροπή σας και στην Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού κάποιες πιο λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τη λογική που ακολουθήσαμε για την εκπόνηση του προπολογισμού. Μιλάμε για ε, ένα προπολογισμό για 1 Πρόκειται για πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων. Έχουμε μία αύξηση 12,8% για τις ε, πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων και ε, έχουμε και αύξηση για τις πιστώσεις πληρωμών πάνω το 2% αυτό εγγράφεται στον ε, αρχικό προγραμματισμό έτσι όπως είχε συμφωνηθεί στις δημοσιονομικές προοπτικές. Όταν αυτές οι δημοσιονομικές ε, προοπτικές συμφωνήθηκαν από δημοσιονομική αρχή προέβλεπαν ε, για τις ε, πιστώσεις στο τομέα ΔΕΗ ένα είδος backloading, δηλαδή σημαντικής ε, αύξησης των πιστώσεων κυρίως προς το τέλος της περίοδου εκτέλεσης και αυτό αντικατοπτρίζει το σχέδιο προϋπολογισμού που σας έχει υποβληθεί. Η αύξηση αυτή θα μας επιτρέψει επίσης ε, να καλύψουμε για το 2011, κατά τη γνώμη μου, τις ε, νέες δημοσιονομικές ε, ανάγκες που θα προκύψουν από την υλοποίηση ή την εκτέλεση του προγράμματος της Οκόλμης, καθώς και του σχεδίου δράσης που μόλις παρουσίασε η Κομισιόν και σας μίλησε και γι' αυτό κυρία Μάστρον προηγουμένως. Αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού έχει επίσης ως συνέπεια την αύξηση του διαθέσιμου περιθωρίου ε, για αυτές τις δημοσιονομικές προοπτικές και το περιθώριο αυτό φτάνει περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την ελάχιστη πρόβλεψη δέσμευσης για τις πιστώσεις για το ΒΙΣ και για το ΣΥΣ 2. Τώρα, ένα θέμα που τέθηκε, μια ερώτηση που τέθηκε και τίθεται όταν διαβάζουμε το προσχέδιο της ε, έκθεσης για την Επιτροπή Προπολογισμών είναι το με ποιο τρόπο ληφθήσαν υπόψη οι ανάγκες των οργανισμών, των agencies. Και εδώ αναγκαστήκαμε να σεβαστούμε την ε, αρχική, τον αρχικό προγραμματισμό που είχαμε συμφωνήσει. Προβλέπονται πιστώσεις για την ε, θέση σε λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου. Αυτές οι πιστώσεις ε, μεταφέρονται όπως είχε συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες και αυτό μας εξηγεί ότι η αύξηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες ε, είναι σχεδόν μηδενική και φυσικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη σημαντική αύξηση των μέσων που έχουν προβληθεί για τα άλλα μεγάλα μέσα αλληλεγγύης για τη διαχείριση μεταναστευτικών πολιτικών. Όμως ε, οι πιστώσεις προβλέπονται πριν τα τέλη του έτους θα πρέπει να επιτρέψουν να υλοποιηθεί, να τεθεί σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου. Προβλέπουμε επίσης πιστώσεις ε, για την μελλοντική ε, για το μελλοντικό οργανισμό διαχείριση των συστημάτων πληροφορική. Ε, έχουμε πιστώσει που μεταφέρονται και είχαν προβλεφθεί για το ΣΥΣ και για το ΒΙΣ, αλλά διατηρούνται τώρα και σε αποθεματικό γιατί πρέπει ακόμη να κάνουμε μια διοργανική συμφωνία για την νομική βάση της δημιουργίας αυτού του οργανισμού. Προβλέπεται μια αύξηση για τις πιστώσεις σε σχέση με τη Eurojust της τάξη ε, του 6% και θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις ε, αποφάσεις που προβληθήκαν πρόσφατα Κυρίως αναφέρουμε στο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο δικαστικών συνδέσμων. Επίσης, ό,τι αφορά την Ευρωπόλ, σεβόμαστε τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, τον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Ίσως ε, στο μέλλον να προκύψει ανάγκη και νέων καθηκόντων, όμως ακόμη δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο σήμερα. Καταρχήν, ε, το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει επί αυτής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας που θα προτείνει η Κομισιόν τον Οκτώβριο και θα αναφέρομαι και πάλι στην παρέμβαση της κυρίας Μάλστρομ. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και εξού και αν χρειαστεί θα προκύψουν και νέα καθήκοντα για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αστυνομίας. Ε, οι πιστώσεις πληρωμών αυξήθηκαν, σας το είπα, η αύξηση αυτή βασίζεται σε μια εκτίμηση των αναγκών μας, επί της ουσίας, αλλά και στην, ε, στο ρυθμό χρήσης ε, των διαθέσιμων πόρων. Και να πω επίσης ότι προσπαθήσαμε να περιορίσουμε το ποσό των δαπανών ε, για τις διοικητικές δαπάνες έτσι ώστε να σεβαστούμε μία πιο επιχειρησιακή ισορροπία. Αυτός ε, είναι ο συλλογισμός που ακολουθήσαμε, Πρόεδρε, σε γενικές γραμμές. Φυσικά να το επιθυμείτε, είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση της Επιτροπής για να απαντήσω σε πιο συγκεκριμένε ερωτήσεις που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε τώρα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα κάνουν σχόλια. Πρώτος ο Σάιμον Μπουσούτιλ. Όχι. Ο κύριος Βαντεν Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για το έγγραφο εργασίας. Είναι σαφές και ξέρουμε πια πώς έχουν τα πράγματα. Κάποιες ερωτήσεις για το 2009. Βλέπω δύο σημεία. Υπήρξε μειωμένη χρήση μέτρων διασφάλισης και εγγύσεων. Κρίμα, λέει η ομάδα μας. Και για τα άλλα προγράμματα υπήρξαν κάποια κονδύλια. Μας δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις για το VIS και SIS. Τώρα για τις προοπτικές το 2011. Στην ομάδα ΕΛΚ χαιρόμαστε πολύ διότι βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός για την ελευθερία, δικαιοσύνη, ασφάλεια θα αυξηθεί. Και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο εμείς στην ομάδα μας. Επίσης, μεγάλη σημασία θα δώσουμε στην εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Αυτό, τα, αυτά τα δεχτήκαμε με πολιτική καλή θέληση. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε όμως και την ε, ύπαρξη κονδυλίων για την εφαρμογή του προγράμματος. Αντιδρούμε θετικά λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Κρίμα που τα κονδύλια του 2009 δεν χρησιμοποιήθηκαν 100% ε, αλλά για το 2011 με χαρά βλέπουμε τις τωρινές εξελίξεις και χαιρόμαστε για τα... Ε, από πριν για την χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Ο κύριος Μπουσουτήλ, τώρα θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω, αλλά σκέφτηκα. Έκλεισε το μικρόφωνο του κύριου Μπουσουτήλ. Εγώ πάντα ήθελα να μιλήσω, αλλά ε, ε, έδωσα το λόγο πρώτα στο σκιώδη. Δεν αλλάζω, μην μην φοβάστε, δεν αλλάζω γνώμη εγώ τόσο γρήγορα. Τώρα, για αυτό που ήθελα να πω. Θέλω να προτείνω κάτι που το έχω ξαναπροτείνει και που αφορά και τη διαδικασία των συζητήσεων και ε, υιοθέτηση της γνωμοδότησης ε, για τον προϋπολογισμό για τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν, ε, είναι δική μας αρμοδιότητα. Εννοώ το εξή. Είναι σαφές ότι οι πολιτικές συζητήσεις στην Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντικές. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος φάκελος είναι ο πιο σημαντικός ίσως από όλους, γιατί χωρίς οικονομικούς πόρους, χωρί χρηματοδότηση, όπω είπε ο κ. Βαντερκάμπ, αν δεν διατεθούν, τι νόημα έχει να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις. Όμως, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποια γνώμη για τον προϋπολογισμό χωρίς να είμαστε σε συνεχή επαφή με τους οργανισμούς που συζητάμε. Θα πρέπει να τους βλέπουμε σε τακτά διαστήματα και να μαθαίνουμε από αυτούς τι σκοπούς έχουν για τον επόμενο χρόνο. Γιατί πώς θα αποφανθούμε για τον προϋπολογισμό του 2011 για τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας αν δεν τους έχουμε δει και δεν έχουμε συζητήσει μαζί τους τι θέλουν να κάνουν του χρόνου. Οπότε πρέπει να καλέσουμε τους υπεύθυνους για, από κάθε οργανισμό που είναι δικής μας αρμοδιότητας να έρθουν εδώ να μας μιλήσουν θα μας πούν τι θέλουν να κάνουν του χρόνου και πάνω σε αυτή τη βάση θα μπορέσουμε και εμείς να έχουμε πιο συνεκτική θέση για τον προϋπολογισμό τους. Και το ίδιο αφορά και τα προγράμματα χρηματοδότησης. Εδώ όμως έχω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, προς την Κομισιόν, η οποία μας είχε υποσχεθεί νωρίτερα κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, ότι θα άρχιζε μια επανεξέταση, η αναθεώρηση των κονδυλίων που δίδονται στα προγράμματα αλληλεγγύης ε, δικής μας αρμοδιότητας και πώς δαπανώνται τα κονδύλια. Πρέπει να γίνει μια λεπτομερής μελέτη από την Κομισιόν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι και εμείς θα διευκολυνθούμε στη λήψη των αποφάσεων όταν θα αποφασίζουμε για τον ε, ε, επόμενο προϋπολογισμό. Η γνωμοδότησή μας θα πάει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, η οποία όμως συνήθως από μας περιμένει να ενημερωθεί για να αποφανθεί οριστικά επί του προϋπολογισμού του επομένου έτους. Οπότε επιμένω κύριε Πρόεδρε, όταν καταπιαστούμε με αυτό το φάκελο θα πρέπει να μπούμε σε μεγάλες λεπτομέρειες και να πάμε σε μεγάλο βάθος και με τους οργανισμούς που μας αφορούν, αλλά και θα πρέπει να μάθουμε πώς τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται από τα προγράμματα χρηματοδότησης στα πλαίσια του κεφαλαίου αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη. Προλίγου είχα ζητήσει στην Επίτροπο κάποια πράγματα, σε μερικά απάντησε, αλλά όχι. Ε, στο ένα συγκεκριμένο ζήτημα και γι' αυτό αποθύνουμε προς την Κομισιόν. Το ε, πρόγραμμα της Οχόλμης και στο σχετικό ψήφισμα προβλέπεται μεταξύ άλλων μια στήριξη αλληλεγγύης κοινωνικής ένταξης των κρατών μελών που έχουν πρόβλημα με την υπερβολική, τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Ε, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά στο ψήφισμα του Νοεμβρίου του 2009 Αναρωτιέμαι λοιπόν, υπάρχουν ικανοί πόροι, υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι, υπάρχουν παράμετροι για την κατανομή αυτών των πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέρη και κάτι ακόμα. Για τους τοξικομανείς όπου για το θέμα αυτό δεν κατορθώσαμε να βάλουμε μια ερώτηση δίχως ψήφισμα στην Ολομέλη σχετικά με την πρόληψη και την ε, επανένταξη τόσο για, την, ε, για τους τοξικομανείς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι λαμβάνοντας υπόψη το 2012 θα ολοκληρωθεί και θα λήξει το πρόγραμμα κατά των ναρκωτικών. Εκεί κ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς, μία ερώτηση προς την Επιτροπή και αν μπορώ έτσι, να έχω κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις. Επειδή στην αρχή αυτή τη θητεία για τον προπολογισμό που ψηφίσαμε για το 2010, θυμάται και ο κύριο που βάλαμε και κάποιες τροπολογίες, αυξήσαμε κάποια ποσά. Ε, και με χαρά πράγματι βλέπω ότι προχωράμε το 2011 σε αύξηση των ε, κονδυλίων για τα θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης. Θα ήθελα να ξέρω για να πορευτούμε έτσι πιο αποτελεσματικά συνέχεια και εμείς στο σώμα και να έχουμε πιο συγκροτημένη άποψη για ποιο λόγο το 2009 κάποια ποσά δεν ξοδεύτηκαν. Φταίνε τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που πήραν. Υπήρξαν γραφειοκρατικά προβλήματα. Υπήρξε κάτι άλλο που θα έπρεπε να έχουμε υπόψη μας για τη συνέχεια και την κατανομή των ποσών. Και δεύτερο, νομίζω κύριε Πρόεδρε και συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, και εγώ ε, βρίσκομαι σε αυτό το σώμα περίπου ένα χρόνο. Πολλοί από εμά νομίζω έχουμε εκλεγεί για πρώτη φορά. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ε, είχαμε στην συνέχεια μια σειρά ακροάσεων με δική σας πρωτοβουλία ή όπως εσείς το κρίνετε καλύτερα, προκειμένου ε, με όλα αυτά τα όργανα που υπάρχουν στη διάθεσή μας και τους οργανισμούς και τα ε, διάφορα προγράμματα, να έχουμε μεγαλύτερη εξοικείωση και να μπορέσουμε επιτελικά να ξέρουμε πώς μπορούμε να έχουμε πιο κατασταλαγμένη άποψη. Ευχαριστώ πολύ. If there are no further comments. Δεν υπάρχουν σχόλια. Τότε είναι η ώρα της Κομισιόν. Κύριε Ντεμπρούβερ. Παρακαλώ να απαντήσετε στα όσα υπόθηκαν. Δηλαδή, επίση κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει ένα σεμινάριο με όλες τις υπηρεσίες και έτσι όχι μόνο θα μπορούμε να προβλέψουμε αλλά και να κρίνουμε τις ε, οικονομικές ανάγκες Κομισιόν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με το ερώτημα για την εκτέλεση του προπορισμού 2009, απαντήσατε εσείς ο ίδιος κύριε Βανερκάμπ για τα μεγάλα προφορικά συστήματα, η εξήγηση είναι προφανής, για τα ιδιαίτερα, ειδικά προγράμματα. Η εξήγηση είναι απλούστατη. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία την χάνουν άμεσης διαχείρισης και προχωράμε σύμφωνα με την κλασική διαδικασία προπολογισμού όπου κάνουμε ε, διαγωνισμούς και αξιολόγηση των προσφορών. Το 2009 αυτήν την άποψη ήταν μια πολύ καλή χρονιά και λάβαμε πολλές προτάσεις περιορισμένου χαρακτήρα και ε, πολλές φορές ε, ε, λοιπούς ε, χαμηλής ποιότητας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μπορέσαμε να δαπανίσουμε τα λεφτά και θελήσαμε να τα δαπανίσουμε όταν θα υπάρχει κατάλληλος λόγος, δηλαδή οι προτάσεις ικανές και αποτελεσματικές. Και κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε σχετικά με τις υπηρεσίες, το πιο προφανές αφορά στην Frontex, ο εκτελεστικός διευθυντής είχε ήδη την ευκαιρία να εκφραστεί ενώπιον της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ε, στην περίπτωση αυτή υπήρξε μια αντιστάθμιση ε, ότι μπορέσαμε να μεταφέρουμε ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την υπηρεσία Frontex τώρα. Σε ό,τι αφορά τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή καταπολέμηση των ε, ναρκωτικών. Ένα ποσό 3 εκατομμυρίων προβλέπεται στο σχέδιο του προπολογισμού για το 2011, δηλαδή ένα ποσό ταυτόσιμο με αυτό που είχε προβλεφθεί και στον προπολογισμό. Στον προπολογισμό λοιπόν 2010, το οποίο εκτελούμε σήμερα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά συνθήκες ε, κράτησης ε, μια γενικότερη σκέψη αναφορικά με τα σωθοδοτικά καταστήματα. Έχετε δίκιο που το τονίζετε αυτόν τον υπερπληθυσμό. Ε, αυτό το και στο πρόγραμμα του Στοχόλμης αλλά και στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Υπάρχει όμως ε, εδώ το ζήτημα αυτού του πιλωτικού προγράμματος, πιλωτικού σχεδίου και χρειάζεται να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Αυτό το σχέδιο, το πιλωτικό, θα πρέπει να χρηματοδοτεί στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια, όπου έχουμε προβλέψει 13.800.000 ευρώ, περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, που ισοδυναμεί με τον προϋπολογισμό που προβλέπονταν ε, για το 2010. Αναφέραμε λοιπόν πως σε αυτό το στάδιο και δεδομένων των αναγγελθέν των προτεραιοτήτων της, από την κυρία Ρέντινγκ που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προγράμματος είναι σαφές λοιπόν ότι τα προγράμματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων και την ε, ιδιωτική σφαίρα και σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο τη εφαρμογή του προγράμματο για του ασυνόδου ανηλίκου, θα αποτελέσουν λοιπόν όλα αυτά προτεραιότητα εντό του προγράμματο του. Τουλάχιστον λοιπόν, εάν κατά τη διάρκεια του έτου υπάρξει συνένεση για το προφίλ αυτού του πολιτικού σχεδίου, τότε σίγουρα θα μπορέσουμε να θέσουμε τις ε, προτεραιότητες ε, στο πλαίσιο του προγραμματισμού. Λοιπόν, τώρα για την αξιολόγηση των ε, προγραμμάτων που τρέχουν, το ερώτηση Μπουζουτήλ για το θέμα του Ταμείου Ελληνικής για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Αυτό το ζήτημα έχει προωθηθεί, αλλά τα αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν από τα τέλη της προσεχούς χρονιάς. Αναφέρομαι εδώ σε μια υπόσχεση την οποία βεβαίωσε και η κυρία Μάλστρομ στην συζήτηση που είχατε κατά διάρκεια του απογεύματος. Προβλέπουμε λοιπόν για το 2011 όχι μόνο μια αναθεώρηση ενδιάμεση των μέσων αλληλεγγύης, αλλά και γενικότερα μια ανακοίνωση για την ενίσχυση της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, εξού και η διαχείριση των ε, μεταναστευτικών ροών. Τώρα, τα οικονομικά μέσα όπως υπάρχουν και όπως γίνει η εκτέλεσή τους μέχρι τώρα αποτελούν ένα στοιχείο της αλληλεγγύης, ένα μέσο αλληλεγγύης. Πρέπει να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, όπως αξιολόγηση προγράμματος επανεγκατάστασης, ε, και, το θέμα της του προγράμματος του Δουβλίνου και νομίζω ότι τα αποτελέσματα ίσως να φτάσουν με κάποια καθυστέρηση, με κάποια για την προπαρασκευή του προϋπολογισμού, την μόνο του προϋπολογισμού από, τις, από την Επιτροπή του 2011. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στα χέρια σας και στα χέρια του Κοινοβουλίου γενικότερα. Λάβαμε υπόψη μας ιδιαίτερα τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των διαφόρων υπηρεσιών για να προτείνουμε το σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο έχετε αναχείρα σήμερα. Το σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό προγραμματισμό αλλά και αυτό το οποίο εκτιμάμε πως αυτό το στάδιο είναι οι ανάγκες αυτών των υπηρεσιών, αλλά αυτό είναι ένα σχέδιο της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή και εσείς είστε μία εκ των δύο. Θα πρέπει να εξετάσετε αυτό το αρχικό σχέδιο. Σας το είπα και προηγούμενα ότι προβλέπετε κάποιο περιθώριο αρκετά γενναιόδωρο, διότι τη τάξη των 5 εκατομμύριων ευρώ, εάν ε, λάβουμε υπόψη την περσινή χρονιά, η αρμόδια για τον προπλησμό αρχή είχε συμφωνήσει στο σύνολό τη για την αύξηση των κονδυλίων που αρχικά προβλέπονταν από την Κομισιόν για την Frontex. Εξάλλου είχαμε βασιστεί σε αυτόν τον προπολογισμό σε ό,τι φορά το προσχέδιο του 2011. Τώρα, αν η Επιτροπή σα θέλει να ε, πράξει το αυτό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη Frontex, αλλά και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπε υπηρεσίε, είναι ε, δικό σα ζήτημα, και σε αρμοδιότητα. Τώρα, το προπολογισμό για τι ε, υπηρεσίε που έχετε αναχείρα ανταποκρίνεται όχι μόνο στον πλανησμό, αλλά και σε μια εκτίμηση των αναγκών του ε, σε σχέση με τι προτεραιότητε στο πρόγραμμα εργασιών του, όπω αυτό έχει αποφασιστεί από τα διάφορα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Νομίζω πως έτσι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα που έτεξαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Δεμπρούερ. Αν δεν Ο κύριος Ντεκάμπ. Μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ότι τα ποσά που είχαν δεσμευτεί για τη Europol ε, ακολουθούν το δημοσιονομικό σχεδιασμό. Της, ποιον σχεδιασμό όμως, του, της Κομισιόν, του Συμβουλίου ή της Europol της ίδιας. Επίσης, άλλη ερώτηση. Τι γίνεται με τους προϋπολογισμούς των οργανισμών. Αυτούς μπορούμε να τους δούμε ή δεν ήθιστε. Εγώ είμαι καινούριο. Αλλά ας πούμε, αν ζητάει ας πούμε 100 ας πούμε η Europol και πάρει 28, ε, τότε τι θα γίνει, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα απαντήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Μιλάμε για το προγραμματισμό που έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο από τη Δημοσιονομική Αρχή. Στι δημοσιονομικέ πολιτικέ που τρέχουν ω το 2013 έχουν προβληθεί προγραμματισμοί για του οργανισμού και αναφέρθηκα σε αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις και αναφερθήκαμε στο Frontex, αυτοί οι προγραμματισμοί ήδη είχαν σκοπίμως υπερβληθεί από τη Δημοσιονομική Αρχή για τη Frontex. Βρισκόμαστε πολύ πιο μακριά από το κατόφλι που είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο του πολιτικού προγραμματισμού, αλλά ε, απλώς ε, βλέπετε ότι η Δημοσιονομική Αρχή αποτεσμοποίησε το διαθέσιμο περιθώριο για να πρικοδοτήσει περισσότερο τη Frontex για την Ευρωπόλ. Μέχρι σήμερα έχουμε ακολουθήσει ε, ένα γραμμικό προγραμματισμό, δεν έχουμε βγει ε, από αυτό. Τώρα, όπως ε, σας είπα για να απαντήσω στην πρώτη σα ερώτηση, θα ήταν δυνατό το γραφείο να θεωρήσει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι αποστολές αυτές, όμως αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί στο μέλλον και δεν θεωρούμε ότι θα ληφθεί απόφαση πριν από τα τέλη του έτους. Έτσι λοιπόν, αν προκύψουν νέες ανάγκες για την Ευρωπόλ, τότε αυτό θα το δούμε κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012, κατά τη διάρκεια αυτών των οικονομικών ετών. Τώρα, για τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις αυτών των οργανισμών και τις προτάσεις της Κομισιόν, να σας πω και πάλι εδώ, Πρόεδρε, ε, συνηθίζεται να καλείτε συχνά τους εκτελεστικούς διευθυντές των οργανισμών ε, για να συζητήσετε εδώ σε αυτές τις επιτροπές, τις κοινοβουλευτικές ε, και πάλι έγκυται στην επιτροπή σας να θέσετε τις ερωτήσεις αυτές στο διάλογο που θα έχετε. Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση για το Frontex, γιατί πολλές φορές αναφέραμε τον οργανισμό. Η Κομισιόν στην πρόταση αναθεώρησης της εντολής του Frontex λέει ότι θα είναι, πρέπει να είναι δυνατόν ο οργανισμός αυτός να αγοράζει ή να μισθώνει ε, κάποια ε, εργαλεία, υποδομή. Έχει γίνει δημοσιονομική πρόβλεψη για αυτή τη δυνατότητα για το 2011 του Κομισιόν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Μπουζουτήλ για την ερώτηση. Αυτό που προβλέπεται στη νομική βάση είναι μια διευκόλυνση αν ψηφιστεί το κείμενο από το συνομοθέτη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο να αποφασίσει, εγκρίνοντας το πρόγραμμα εργασία του οργανισμού, αν ναι ή όχι θα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, αν θέλει να αγοράσει εξοπλισμό, τι είδου εξοπλισμό, αν επιθυμεί να προβεί σε μίσθωση, γιατί και αυτό προβλέπεται από τη νομική βάση έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή θα γίνει εξελόγηση του δημοσιονομικού κόστους στον ε, χρηματοοικονομικό προγραμματισμό του οργανισμού. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε στάδια ε, θα πρέπει καταρχήν να συμφωνήσουμε μέσω της απόφασης για να δούμε αν θα αναλάβει αυτές τις αρμοδιότητες ε, η Frontex. Αν είναι θετική απάντηση τότε η Frontex θα είναι αρμόδια για να αποφασίσει αν θέλει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή και ω πιο ύψο, ω πιο ποσό και τότε θα προβούμε στις απαραίτητε δημοσιονομικές προσαρμογές. Ε, ήδη ο μηχανισμός αυτός έχει αναπτυχθεί στο δελτίο το οποίο το βλέπετε ω παράρτημα στην πρόταση. Ευχαριστώ. Νομίζω λοιπόν τώρα ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γιατί πραγματικά έχουμε καθυστερήσει και έχουμε κάποια ακόμα σημεία που πρέπει να εξετάσουμε και έχουμε μόνο 20 λεπτά πριν τη συνεδρία των συντονιστών. Ξέρετε τώρα ποια είναι η επίσημη απόφαση της δηλαδή ΛΥΠΗ. Θα πρέπει οι τροπολογίες να ετοιμαστούν πριν από το καλοκαίρι, προκειμένου να θετηθούν από τη ΛΥΜΠΕ αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι λοιπόν, ε, σκοπεύεται να παρουσιαστεί ένα δεύτερο έγγραφο εργασία με ανάλυση και προτάσεις στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αν συμφωνείτε, τότε προχωρούμε στο επόμενο σημείο το υπερθυμόν 7, κυβέρνηση του διαδικτύου, τα επόμενα βήματα. Έχουμε τον κύριο Λαμπρινίδη, ο οποίος είναι συντάκτης της νομοδότησης, αν θέλετε. Παρουσιάστε μας ε, το σχέδιο γνωμοδότησής σας και να σας πω τροπολογία για ε, η, συγγνώμη, για την κατάθεση τροπολογιών ε, θα πρέπει να τεθεί στις 14 Μαΐου, πέμπτη με το μεσημέρι. Όχι, Παρασκευή διορθώνει ο μίλητη. Παρασκευή μεσημέρι στις 12. Κύριε Λαμπρινίδη. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι, αναφέρεται στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο κύριος Φρανσίσκο Βάγνερ είναι ο εισηγητής και αφορά το μέλλον της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Γενική έκθεση πρέπει να πω που επικεντρώνει σε θέματα όπως το ICANN, που είναι μη κυβερνητική, ε, ε, ε, κερδοσκοπική οργάνωση ε, και αν μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που μπορεί κανείς να προτείνει για την καλύτερη διακυβέρνηση του διαδικτύου μέσω του ICANN, αυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης αλλά επειδή η γνωμοδότησή μα ως ΛΥΜΠΕ πρέπει να επικεντρώνεται στα δικά μα τα θέματα κυρίως, θα σημειώσετε και τονίζω τι πρώτε τρεις παραγράφους κυρίως. Αυτά θα πρέπει να αναφέρει η γνωμοδότησή μα στην ε, πρότασή της για την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σε προηγούμενες εκθέσεις και στη δική μου είχαμε πει ότι θέλουμε όλες οι συζητήσεις ε, στο μέλλον ε, για το θέμα αυτό της διακυβέρνησης να συμπεριλαμβάνουν όλους τους εμπλεκομένους ε, σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Θέλουμε να διασφαλιστεί ότι θα, θα προστατεύεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε θεμελιώδες δικαίωμα. Επίσης ε, θα αντιμετωπίσουμε τη διπλή πρόκληση της ηλεκτρονικ... του ηλεκτρονικού του δημοκρατικού αποκλεισμού. Το δεύτερο θα πρέπει να σχεδιάσουμε διασφαλίσεις ε, της ιδιωτικής σφαίρας ε, παγκοσμίως και η εναρμόνιση πολλές φορές συζητείται από κάτω προς τα πάνω. Θα πρέπει λοιπόν αρχικά να έχουμε δει αυτά τα θέματα, να τα έχουμε προβλέψει. Επίσης θέματα επιτήρησης, ελεγχόμενης λογοκρισίας από δρόντες, ιδιώτες και δημοσίους που θα πρέπει να περιορίζεται στο απόλυτο ελάχιστο που απαιτείται και στο τρίτο σημείο Αναφέρομαι στο χάρτη δικαιωμάτων ή τον ε, νόμο ε, των δικαιωμάτων του διαδικτύου στην έρευνα και την ανάπτυξη ως διαδικασίες. Ε, δεν είναι και τίποτε το, το καταπληκτικό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνουμε στο, να συμπεριληφθούν αυτά τα θέματα γιατί ως Επιτροπή κατά το παρελθόν θεωρούσαμε ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Λαμπρινίδη που μας παρουσιάσατε το σχέδιο γνωμοδότησης και τώρα οι συνάδελφοι. Ο κύριος Φως έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η σημασία του διαδικτύου αναμφίβολα αυξάνει και το μεταξύ έφτασε σε ένα επίπεδο που επηρεάζει ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Και η σημασία του αυξήθηκε και στα θέματα της παιδείας, της ενημέρωσης, της επικοινωνίας γενικότερα. Άπτεται επίσης εν μέρη και θεμάτων ασφάλειας. Και σε τελευταία ανάλυση πρέπει να πούμε ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσον του μέλλοντος. Η σημασία του έχει αυξηθεί τόσο πολύ εντωμεταξύ που θεωρείται ως υποδομή του, του σημερινού μας κόσμου και αν θέλετε συγκρίνεται με άλλες υποδομές που κατά κανόνα ρυθμίζονται από δημόσιους φορείς. Έτσι το διαδίκτυο πολύ περισσότερο θα πρέπει να αξιολογηθεί ε, στον πύχη του δημοσίου συμφέροντος και θα πρέπει γι' αυτό να έχουμε αποτελεσματική διακυβέρνησή του, διοίκησή του. Πώς μπορούμε λοιπόν το παρόν στάτους του ICAN να το αναβαθμίσουμε και να προσπαθήσουμε να το επηρεάσουμε. Ε, και πέραν τούτου υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι το ίντερνετ θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις επιμέρους απαιτήσει. Ε, ο αυτοπροσδιορισμός του είναι σημαντικός εδώ και πρέπει να θέσουμε και το θέμα της ασφάλειας. Πώς θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα πλαίσιο ρύθμισης του διαδικτύου που θα ισορροπεί μεταξύ ελευθερίας του διαδικτύου, που είναι καλό πράγμα, Παράλληλα όμως θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο που θα διασφαλίζει θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του καθενός που, μπαίνει στο διαδίκτυο. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ελευθερίες ε, ποτέ δεν είναι αέναες και ανεφορίων και τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα των άλλων. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στα σημεία 6 και 7 της έκθεσης ως παράδειγμα. Βεβαίως θεωρώ ότι χρειάζεται τρόπον την άμια επιτήρηση, επίβλεψη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκληματικέ δραστηριότητες. Γι' αυτό δεν συμφωνώ τόσο πολύ με την επιλογή των λέξεων στο σημείο 6 που, και, ε, για τα διάφορα συμφέροντα. Και επίσης ε, να περιορίσουμε ένα ε, ε, ελάχιστο μέτρο όταν πρόκειται για ανηλίκους. Και αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί δεν νομίζω ότι οι ανήλικοι θα πρέπει κατ' ελάχιστο να προστατεύονται, αλλά μάλλον κατά μέγιστον ή περιεκτικότερα τέλο πάντων. Ευχαριστώ κύριος Γιακολίνο. Πολύ σύντομα το ζήτημα του ίντερνετ ε, φυσικά ενέχει μια σειρά από αξιολογήσεις. Ε, συμφωνώ με ένα μεγάλο κομμάτι της ε, έκθεσης όπως την εξεντάξει ο συγητής. Ορισμένες προτάσεις δεν είναι... Είναι μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια πιο υπεύθυνη συμμετοχή των, του ιδιωτικού και του δημοσίου κλάδου. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση περί αυτού όλοι αναγνωρίζουμε ότι το ίντερνετ μπορεί να οδηγήσει σε εξαρτήσεις σημαντικές. Και εδώ υπάρχει το θέμα της προστασίας ε, των πλέον ευάλωτων που δεν είναι μόνο τα παιδιά. Ε, Παραδείγματος χάρη, τα, ο τζόγος μέσω ίντερνετ, ε, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσουν ε, είναι κάτι το οποίο έχει επανειλημμένα εξετάσει στο Κοινοβούλιο, αλλά προφανώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των ευάλωτων προσώπων και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση του ζητητή. Ευχαριστώ τον Μπρόντσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το διαδίκτυο ε, εξισορροπεί ε, τις πολιτικές δυνάμεις που, δηλαδή καπιταλιστικά ισχυρούς και άλλους που παραγνωρίζονται. Ε, βεβαίως στο διαδίκτυο, στο, μέσα από το διαδίκτυο γίνονται και εγκληματικές δραστηριότητες. Σίγουρα πρέπει αυτές οι δραστηριότητες να περιστέλλονται, αλλά δεν πρέπει η διακυβέρνηση να ε, λογοκρίνει ακαδημαϊκές απόψεις. Ε, αυτό γινόταν ε, από τυραννικά καθεστώτα στο παρελθόν και ας μη μας ξεγελάει η επίφαση της δημοκρατικής τους γλώσσας σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Σταβάρης. Απλώς να πω ότι γενικά υποστηρίζουμε τη γνωμοδότηση αυτή Φαίνεται ότι δίνει την ορθή έμφαση στην πολυμερή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του διαδικτύου, κυρίω σε φορέ όπω το ICAN. Και περιλαμβάνονται και κάποιε ενδιαφέρουσε ιδέε για την ηλεκτρονική δημοκρατία. Και ο Σκιώδη ε, εισηγητή ε, δεν μπορεί να παρευρίσκεται εδώ, αλλά μα είπε να εκφράσουμε την υποστήριξή του και θα παρουσιάσει και κάποιε ιδέε στο μέλλον. Αλλά γενικά εμεί υποστηρίζουμε την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, πάλι σας δώσουμε το λόγο, κύριε Λαμπρινίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι είναι όλοι ενθουσιώδεις, γιατί πράγματι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν αναφέρεται αυτή η γνωμοδότηση στη γενική φιλοσοφία του διαδικτύου, απλώς τονίζει την πτυχή της διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά τις παραγράφους που αναφέρατε, πράγματι, Αναφέρεται στο σχεδίο έκθεσης ε, τη Επιτροπή βιομηχανία ε, και όχι στη δική μου νομοδότηση, παράγραφα 6 και 7. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν αφορούν το δικό μου έγγραφο. Το κείμενο της Επιτροπής ΙΤΡΕ φυσικά μπορεί να αλλάξει στα σημεία αυτά. Εγώ αναφέρθηκα σε κάποια από τα σημεία αυτά, αλλά χρησιμοποίησα τη γενική διατύπωση που χρησιμοποιούμε πάντα, δηλαδή δεν ε, θέλουμε λογοκρισία, έλεγχο, εποπτεία χωρίς να χρειάζεται. Και ε, επίσης ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον οποιαδήποτε τέτοια μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα και αναλογικά. Πάντοτε αυτό έχουμε δηλώσει. Έτσι λοιπόν εκτιμώ τα σχόλια που ακούστηκαν. Αλλά όσοι αναφέρθηκαν απευθεία στην γνωμοδότησή μου, ευχαριστώ να μου στείλετε τροπολογίες. Αν ε, θέλετε μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το γραφείο μου ή για μένα απευθεία τις επόμενες ημέρες και ευχαριστώ να συζητήσουμε τα σχόλιά σας. εγκαίρω προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορώ να τα υποστηρίξω πλήρω. Αλλά φυσικά αν δεν προλαβαίνετε, τότε ευχαρίστω ε, να μου τα στείλετε και να προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λαμπρινίδη και όλους σας ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας. Χαίρομαι που καλύψαμε τόσο μαλά αυτό το σημείο στην στη διάταξη. Να σας υπενθυμίσω ότι οι προθεσμοί για την κατάθεση τροπολογιών είναι Παρασκευή 14 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 8 να σας πω ότι τα σημεία 9 και 10 έχουν αναβληθεί. Έτσι λοιπόν, αυτό θα είναι το τελευταίο σημείο στην ημερησία διάταξη πριν από τη συνεδρία των συντονιστών. Αυτό το σημείο αφορά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία και Νορβηγία για την εφαρμογή διατάξεων της απόφαση του Συμβουλίου 2008 615 ΔΕΗ και της απόφασης του Συμβουλίου 2008 κάθετος 616. Εδώ θα ακούσουμε τον συγκεκριτή, τον κύριο Βουσουτήλ. αλλά να σας υπενθυμίσω ότι στη συνάντησή μας στις 7 Απριλίου Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη συμφωνία. Μας ε, ενημέρωσαν και για την κατάσταση της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι η για την κατάσταση τροπολογιών τίθεται επίσης στις 14 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η συμφωνία δεν μπορούσε να τροποποιηθεί. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον ιστορικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι τροπολογίε θα μπορούσαν να στελούν ε, στο σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος, αλλά μόνο αν αναφέρονται σε διαδικαστικές πτυχε. Έτσι λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα τον συγκητή, τον κύριο Μπουσουτήλ, και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στου συνάδελφου Κύριε Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Για να κερδίσουμε κάποιο χρόνο, θα είμαι πολύ σύντομο. Είναι τεχνικό το ζήτημα αυτό και πρέπει να πούμε ναι ή όχι στην ε, επέκταση της συμφωνίας στην Ορβηγία και στην Ισλανδία την ε, εφαρμογή διατάξεων μια συμφωνίας που ήδη εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη διασυνορική συνεργασία, την καταπολέμηση της τρομοκρατία και την καταπολεμήση του διασυνοριακού εγκλήματο. Όπως είπατε, είχαμε μια παρόμοια ανταλλαγή απόψεων. Είπαμε ότι αυτό είναι σημαντικό για αυτές τις δύο χώρε, αλλά σημαντικό και για εμά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεργαστούμε με την Νορβηγία και την Ισλανδία για την καταπολέμηση του εγκλήματο και της τρομοκρατία. Όπω ξέρετε, από τη θέση της εφαρμογή της Αγώνας έχουμε την αρμοδιότητα της συνένεσης για το φακελό Έτσι λοιπόν έχουμε την εξουσία να πούμε ναι ή όχι. Και μόνο τότε θα μπορέσει να εγκρίθει αυτή η συμφωνία και να τη ισχύ. Έτσι λοιπόν, η συστασία μου είναι πολύ απλή. Εγώ συστήνω να πούμε ναι σε αυτή τη συμφωνία γιατί είναι καλή και σημαντική και για την Ισλανδία και την Νορβηγία, αλλά και για μας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μπουσουτή. Η Κομισιόν ή η Προεδρία του Συμβουλίου ή κάποιος άλλος συνάδελφος θέλουν να σχολιάσουν. Θέλετε να σχολιάσετε μήπως αυτή την πρόταση του κύριου Μπουσούτιλ για θετική απάντηση. Αν όχι, να προχωρήσουμε στα διάφορα.